Πάμε λοιπόν, έχουμε αρκετούς ε, βουλευτέ, ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι τα θέματα των δημοσίων οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και ο εισηγητή είναι ο Αλφέρντο Παλώνη, στον οποίο δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους ε, συναδέλφους και τους κοιόδης εισηγητές για την ε, πολύ σημαντική συμβολή τους κατά τη σύνταξη της έκθεσης αυτής. 126 είναι οι τροπολογίες και νομίζω ότι στις τροπολογίες αυτές τελικά είχαμε μια πολύ σημαντική πολιτισμική θα έλεγα συμβολή και είμαι σίγουρος ότι οι τροπολογίες αυτές θα καταλήξουν σε πολύ καλούς ε, συμβιβασμούς. Συμβιβασμοί που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε μια ψηφοφορία κατά την οποία θα έχουμε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης αυτής. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε, κυρία Πρόεδρε, είναι γνωστή. Στις 12 Νοεμβρίου, στις 6.30, θα συναντηθώ με όλους τους κοιόδης ηγητές, προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές λύσεις, σε μια κοινή συνένεση, Μέσω μιας εργασίας προσπαθώ κάπως να διαμορφώσω αυτή τη στιγμή και στις 19 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε στο Στρασβούργο. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω σε αυτή τη φάση είναι ότι προσπαθώ να αξιολογήσω κάποιες τροπολογίες στις οποίες ουσιαστικά θα έχουμε δύο διαφορετικές σχολές. Υπάρχουν βέβαια οι δύο αυτές σχολές που θέλουν την οικονομική ανάπτυξη στα κράτη-μέλη, αλλά μια σχολή θεωρεί ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το six-pack, με το του pack ότι μάλλον οι νομοθεσίες αυτές για το six-pack δεν μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και δεν επιφέρουν πολύ σημαντικά ωφέλη, ενώ υπάρχει η άλλη σχολή που λέει ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς σίγουρα, αλλά θα πρέπει επίσης να καταφέρουμε να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη κάνοντας τις απαραίτητες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και κάνοντας παράλληλα και πολύ σημαντικές επενδύσεις όσον αφορά την καινοτομία και όσον αφορά την κατάρτιση, την εκπαίδευση. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, θα υπάρχει μια κάποια αντιπαράθεση αλλά θα πρέπει να έχουμε μια παρότητη, απαραίτητη διανοητική ειλικρίνεια, αν θέλετε. Πρόκειται λοιπόν για δύο σχολές που όμως έχουν θέσει έναν κοινό στόχο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξής, ότι κανείς τελικά δεν έχει την απόλυτη αλήθεια. Θα πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε κάποια κοινά σημεία όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης, ιδίως σε μια στιγμή η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ήπειρά μας μια στιγμή όπου υπάρχουν πάρα πολλές ε, αντιευρωπαϊκές λαϊκιστικές τάσεις στις χώρες μας. Ακόμα και στη δική μου τη χώρα γίνεται μια προσπάθεια να προθωθεί μια δημαγωγική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει πραγματικά να θέσουμε ψηλά τον πύχη και να καταφέρουμε να κάνουμε μια αντιπαράθεση ιδεών γόνιμη η οποία θα λειτουργήσει υπέρ των πολιτών. Στις 12 λοιπόν Νοεμβρίου θα ξεκινήσουμε τη συνάντηση αυτή, τη συζήτηση αυτή, χωρίς να είμαι καθόλου προκατηλημένος, με απόλυτη αντικειμενικότητα. Οι περισσότερες άλλες τροπολογίες που έχουν ήδη κατατεθεί συμβάλλουν στο να βελτιωθεί το κείμενο. Βελτιώνεται λοιπόν το κείμενο όχι με τρόπο μονομερή, αλλά με τρόπο πολύπλοκο, πολύπλευρο. Έτσι λοιπόν στις 19 Νοεμβρίου στις 6.30 θα διοργανώσω αυτή τη συνάντηση κυρία Πρόεδρε προσπαθώντας να πετύχω την καλύτερη δυνατή συμφωνία όσον αφορά τις τροπολογίες αυτές. Ε, Merci, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. <clears throat> Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Σιγητά, μετά από την ε, τελευταία ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στην Επιτροπή μας για την εκθεσή σας. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει για το κείμενο αυτό και είχα την ευκαιρία να σας πω ότι βέβαια διατρέχεται από κάποιο δογματισμό, αλλά με ένα πιο επικοδομητικό πνεύμα από ό,τι στο παρελθόν καταλήξαμε στην κατάθεση μια σειρά τροπολογιών που έχουν σαν στόχο να επαναπροσανατολίσουν λιγάκι το κείμενο αυτό, ώστε να βρίσκεται πιο πολύ ε, σε συμφωνία με την οικονομική κατάσταση και συγκυρία στην Ευρώπη. Η δική μου πολιτική ομάδα δεν είναι βέβαια η μόνη η οποία αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες με, την, ε, με τις διατυπώσεις σας και οι 126 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για μία έκθεση τριών σελίδων καταδεικνύουν ότι υπάρχει ένα τέτοιο πνεύμα. Πριν ξεκινήσουμε όμως συζήτηση για τις τροπολογίες, πρέπει να εκφράσω την λύπη μου για, λύπη μου για το γεγονός ότι εσείς δεν έχετε δείξει κατά την σύνταξη του πρώτου σχεδίου έκθεσης ένα πνεύμα αντίστοιχης συνεργασίας. Σε ένα συναφές έγγραφο εργασίας εμείς θεωρήσαμε ότι επειδή δεν υπήρχε μια επαρκή συνεργασία, Ορισμένοι από εμά αναγκαστήκαμε να απειλήσουμε με την συνολική του απόρριψη. Βλέπω ότι εσείς τώρα όμως κάνετε μία προσπάθεια για συνεργασία, αλλά σας προσκαλώ να είστε ακόμα πιο επικοδομητικό στο μέλλον για τα θέματα αυτά. Για τώρα στην ουσία του θέματος. Οι 26 τροπολογίες που έχω καταθέσει εγώ προσωπικά υπενθυμίσουν τις οικονομικές εξελίξεις και τις πολιτικές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα πρόσφατα από την, ε, ε, από την δημοσίευση της αρχικής έκθεσης του 2011 και του 2012. Όπως ξέρετε έχει αυξηθεί η ανεργία και έχει υπάρξει ύφεση σε πολλές χώρες της ζώνης του ευρώ. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί ιδίω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που καταδεικνύουν τον υφεσιακό χαρακτήρα της πολιτικής λιτότητος και επίσης υπάρχει και μία ανακατεύθυνση της ε, οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα γνωρίσει. Πώς θα μπορέσουμε να αναλύσουμε τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να λάβουμε υπόψη τον αντίκτυπο που έχουν στον οικονομικό στίβο και όταν βλέπουμε ότι η Ευρώπη αρχίζει πια να ξεφεύγει από την ψευδέστηση ότι η λιτότητα θα λύσει τα προβλήματα. Όταν λέτε ότι η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη, ξεχνάτε να πείτε ότι και η ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για την εξυγίανση των δημοσιονομικών λέτε ότι χρειάζεται να υπάρξει συγκράτηση των δαπανών για να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση. Δυστυχώ οι μελέτε του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου ανα, ε, επαναυπολογίζουν τον πολλαπλασιαστή των δημοσίων δαπανών και ανασκευάζουν αυτή τη θέση. Επίση, έχουμε αναφερθεί ιδιαίτερα στα θέματα της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ ε, και της ανάγκης να υπάρχει μια τέτοια διακυβέρνηση εκ των προτέρων και όχι μονάχα εκ των υστέρων. Πιστεύω παρόλα αυτά ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμβαστική λύση σε σχέση με το σχέδιο έκθεσή σα, αλλά θα πρέπει να εργαστείτε κι εσεί για να υπάρχει μια καλύτερη προσέγγιση των θέσεων και περιμένω λοιπόν τη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιον από του φιλελεύθερου. Ο Σφεν νομίζω ότι ε, γίνεται πατέρας ε, όπου να είναι, οπότε γι' αυτό το λόγο δεν είναι παρόν. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Βενέτ. Εγώ θα ήθελα απλώς να σας πω ότι ο Σβέν είναι υποχρεωμένος να μείνει στη Γερμανία και δεν μπορεί να λάβει το λόγο και ο άλλος συνάδελφός μου από την ομάδα των Πρασίνων δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα αλλά θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον εισηγητή ότι και οι δύο θα συνεχίσουν να παρακολουθούν το θέμα αυτό και είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί του και λυπάμαι που δεν μπορώ εγώ να εκφέρω γνώμη επί της ουσίας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ο Ντέρκ. Και εγώ ως νέος πατέρας ξέρω πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα αυτά. Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του. Στην ε, τωρινή μορφή της έκθεσής του, η συντηρητική και μεταρρυθμιστική ομάδα μπορεί να την υποστηρίξει πλήρως. Τονίζουμε ότι η εξυγίανση των δημοσιονομικών είναι μια αναγκαιότητα στις χώρες του ευρώ. Θα πρέπει το εξάπτυχο, το six-pack, να εφαρμοστεί πλήρω. Επίση, υποστηρίζουμε αυτά που λέει ο εισηγητή για μεταρρυθμίσει οι οποίε θα πρέπει να οδηγήσουν σε ανάπτυξη, να μειωθούν οι δημόσιε δαπάνε και η φορολογία και να εξυγχρονιστούν τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Βλέποντα τι τροπολογίε που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι, έχω διαπιστώσει ότι πολλέ πολιτικέ ομάδε αντιμετωπίζουν αυτή την έκθεση σαν να είναι κατάλογο ονείων και επιθυμιών. Οι τροπολογίε που θέλουν να προσθέσουν ξεκινούν από τα ευρωομόλογα και φτάνουν μέχρι την εναρμόνιση του φόρου επιχειρήσεων. Υπάρχουν εκκλήσεις επίσης για περισσότερους ίδιους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν αυτό να είναι αυτός σκοπός και τρόπος να μειωθούν οι μακροοικονομικές και οικονομικές ανισομέρειες. Υπάρχει ακόμα και μια τροπολογία για τη βελτίωση των πολιτικών στον εργασιακό χώρο με τη μείωση των ωρών εργασίας. Είναι περιττό να σας πω ότι όλες αυτές οι τροπολογίες δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο και φυσικά δεν είναι αποδεκτές από τη δική μου ομάδα. Γιατί θα οδηγούσαν σε λιγότερη ανταγωνιστικότητα, λιγότερη ε, ανάπτυξη, λιγότερη απασχόληση. Όλα αυτά είναι ένας φαντασιακός χώρος, αλλά τα αρνητικά του αποτελέσματα θα είναι συντριπτικά. Γι' αυτό το λόγο, κυρία Πρόεδρε, θέλω να ενθαρρύνω τον εισηγητή να παραμείνει στο αρχικό πνεύμα της έκθεσής του, και να προσβλέψει σε μια θετική συνεργασία για τις τροπολογίες συμβασμού. Ευχαριστώ. Ο Τόμας Χέντελ από την Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτά που είπε ο προελής σας. Ε, βέβαια δεν θα τα πω αυτή τη στιγμή γιατί θα υπάρξει η συζήτηση των ε, σκιωδών και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ στον εισηγητή. Και θέλω να πω το εξής. Ε, από τις παρατηρήσεις που έκανε προκύπτει ένας τέτοιος προσανατολισμός που οδηγεί στο είτε το ένα είτε το άλλο, είτε μαύρο είτε άσπρο. Εγώ όμως νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ, σε αυτή την υπόθεση, δεν είναι όλα μαύρο-άσπρο για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία όσον αφορά τη θέση της δικής μας της πολιτικής ομάδας, θέλω να πω ότι η εξυγίανση του προπολογισμού είναι σαφώς και πολύ σημαντική και κανείς ε, δεν τάστε υπέρ του να διασπαθίζονται κονδύλια και να προκύπτουν υπέρογκα χρέη. Δεν πρόκειται περί αυτού. Νομίζω όμως ότι από τις ε, τροπολογίες ε, που έχουν κατατεθεί προκύπτουν πολλές θέσεις που δείχνουν ότι το θέμα δεν είναι μόνο να εξετάζουμε με τις δαπάνες αλλά και τα έσοδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, θέλει να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να αναθεωρηθεί εκ βάθρων η πολιτική λιτότητα των τελευταίων τεσσάρων ετών. Σε μια τέτοια λοιπόν έκτηση ε, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για επιζήμιες ε, επιπτώσεις των εσόδων ε, βλέποντας το τι γίνεται στην Ευρώπη. Έχουμε 36 δισεκατομμύρια ιδιωτικές καταθέσεις στην Ευρώπη. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ε, όσον αφορά το θέμα αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά την ανακατανομή των εσόδων και αυτό να προκύψει σε μια αντίστοιχη έκθεση. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να αναφέρεται και η κοινή αγορά στις χώρες που έχουν πλεονάσματα και επίσης ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μία μακροχρόνια ισορροπία ανάμεσα στις πλεονασματικές και τις ελληματικές χώρες. Το θέμα του επίπεδου φορολογίας στην Ευρώπη πρέπει να συζητηθεί. Όποιος λοιπόν επιθυμεί ο ευρωσκεπτικισμός να μην αυξηθεί σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποιος το επιθυμεί αυτό, δεν μπορεί να ε, συνεχίσει ε, την πολιτική εις των χαμηλόμισθων, αλλά πρέπει να αναζητήσει μια ισορροπία ισορροπημένη κοινωνική πολιτική. Δηλαδή οι πιο πλούσιοι να φέρουν μεγαλύτερο βάρος και αυτό είναι το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε στη συζήτηση των σκιωδών συζητών. Και αν γίνει αυτό νομίζω ότι θα είναι μια πολύ λογική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ο Ζαν Πολ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την εργασία που έχει κάνει. Συγγνώμη για το μικρόφωνο. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τον εισηγητή μας για την εργασία που έχει κάνει, τι προσπάθειες που έχει καταβάλει και θα ήθελα κι εγώ, εφόσον δεν υπάρχει εδώ πέρα πάρα πολλοί κόσμος, να αντιδράσω στα όσα είπε ο συνάδελφο Λίν. Είναι πολύ νέο ουσιαστικά για να έχει γνωρίσει το 1968 και νομίζω ότι σηματοδότησε εποχή η περίοδος αυτή. Οι φίλοι του Κον Μπεντή την εποχή εκείνη λέγανε λόγια όχι πράξεις. Νομίζω όμως ότι α, οι α, ουσιαστικά έχουν τελικά υιοθετήσει πλέον πλήρως τη στάση αυτή καθότι ακούμε μόνο λόγια και περιμένουμε να δούμε στην πράξη τι τελικά θα γίνει. Αναλύοντας λοιπόν την οικονομική κρίση, συντοποιούμε ότι ε, μέσα σε μερικούς μήνες, μολονότι δεν έχει συμβεί τίποτα ουσιαστικό, οι αναλύσεις ξαφνικά τροποποιούνται. Για τους ε, οικονομολόγους βέβαια μπορούν να υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις, όσο και οι οικονομολόγοι τελικά, αρκεί να μην ε, έρχονται μία σε αντίθεση με την άλλη. Έχω ασχοληθεί επίσης με την οικονομία, όπως και με την νομική, ενδεχομένως αυτό να με βοηθάει στην ανάλυση μου. Βλέπουμε επίσης ότι αλλάζουν οι αναλύσεις, αναλάζουν οι θεωρητικές αντιμετωπίσεις και έχουμε περάσει από μια μεγάλη κρίση, όπως λέμε στη Γαλλία, προς μια κρίση από την οποία αρχίζουμε σιγά σιγά να βγαίνουμε, υποτίθεται. Εγώ δεν βλέπω όμως κάποια αλλαγή και δεν βλέπω ότι υπάρχουν χώρες, ιδίω οι πιο ευάλωτε χώρε, οι οποίε καταφέρουν να βγουν από την κρίση. Λέμε ότι χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη. Πολύ ωραία, αλλά πώ θα επιτευχθεί αυτή η οικονομική ανάπτυξη. Ο Λίν μα είπε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την οικονομική αυτή ανάπτυξη. Από την άλλη όμως χρειαζόμαστε την οικονομική ανάπτυξη προκειμένου οι οικονομίες μας να είναι πιο βιώσιμες. Το πρόβλημα είναι ότι όταν το χρέος είναι πάρα πολύ μεγάλο, όταν αντιμετωπίζουμε οικονομικές δυσκολίες, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να εξισορροπούμε τα πράγματα. Αυτό πρέπει να γίνει προφανώ με ισότητα και δικαιοσύνη και σαφώ θα πρέπει να κατακρίνουμε τα όσα γίνονται στι χώρες οι οποίες βρίσκονται σε πολύ δυσμενή κατάσταση. Λαμβάνονται κάποιε ανεύθυνε αποφάσει οι οποίες ε, δεν λαμβάνουν υπόψη τους την πραγματική ανάλυση των πραγμάτων. Αναφέρομαι για παράδειγμα στην Ελλάδα, όπου το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει μέτρα πολύ πιο δύσκολα, τα οποία δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν ακριβώς επειδή είναι αβάστακτα. Είναι πάρα πολύ θετικό λοιπόν ότι ο εισηγητή μα αναφέρεται στα ζητήματα αυτά. Πιστεύω ότι σαφώ θα πρέπει να βρούμε κάποιε συμβαστικέ λύσει. Ξέρω όμω και για το ΛΙΝ ο συμβασμό δεν θα είναι απλώ να ευθυγραμμιστούμε με την αντιμετώπιση των άλλων, δεν θα είναι αυτό ο συμβασμό. Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε τι απόψει μα, προκειμένου η εργασία που κάνουμε εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια σύντομη έκθεση, να είναι σε θέση να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα. Και όπω είπε και ο συνάδελφο Έπινγκ, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να Έχουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα στην έκθεση αυτή, αλλά να εστιαστούμε σε δύο-τρία σημαντικά πράγματα, προκειμένου να καταφέρουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο άλλο που θα θέλει το λόγο, κύριε Ποδηματά. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, Σάρον. Uh, να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις, εφόσον κάνουμε εδώ πέρα μια συζήτηση. Και να βασιστώ λίγο και στις παρατηρήσεις uh, του Ζαν Πολ. Βρισκόμαστε λίγες ώρες, uh, λίγες ώρες προτού διεξαχθεί μια πολύ δύσκολη ψηφοφορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για κάποια πολύ σκληρά δημοσιονομικά μέτρα στα πλαίσια μιας ύφεση η οποία έχει ξεπεράσει το 6,3% και ένα ποσοστό ανεργίας το οποίο έχει ξεπεράσει το 23%. Δεδομένης λοιπόν αυτής της χρονικής στιγμής θεωρώ ότι η έκθεση του κυρίου Παλώνε μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση όσον αφορά τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να υιοθετηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήδη εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω στι χώρε που αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα κρίση. Θα ήθελα καταρχάς και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας για την εργασία που έχει κάνει, για το σχέδιο αυτοέκθεσης και θα ήθελα απλώς να υπογραμμίσω ότι ε, πιστεύω ότι το ψήφισμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι πιο ισορροπημένο και πιο ρεαλιστικό. Σε συνέχεια, τον όσον είπε ο συνάδελφος Λίαμ, πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες αυτές τις νέες πληροφορίες τις οποίες έχουμε πλέον στα χέρια μας, όπως για παράδειγμα την παγκόσμια αναγνώριση η οποία περιλαμβάνεται καθώς επίσης στις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν έχουμε εκτιμήσει ακριβώς τα μέτρα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, καθώς επίσης και αυτό το οποίο ονομάζουμε δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να δούμε πώς τα μέτρα αυτά εξυγίανσης επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη δημοσιονομική ισορροπία στα κράτη-μέλη και πώς αυτό σχετίζεται με τη βιωσιμότητα του χρέους καθώς επίσης και με τη δυνατότητα ίσπραξης των φόρων. Οι πρόσφατες αποφάσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ζήτησαν ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πιο διαρθρωμένη μεταρρύθμιση, μια δημοσιονομική εξυγίανση και προσαρμογή, η οποία θα είναι πιο φιλική και η οποία θα συνάδει τελικά με την Ευρωπαϊκή 2020. Νομίζω ότι και η στρατηγική αυτή, η στοιχεία της στρατηγικής αυτής θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο ψήφισμά μας και για να μην με παρανοήσετε πιστεύω ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε τις ιδιαιτερότητες μεμονωμένων κρατών μελών, ιδιαιτερότητες που οδηγούν σε εντελώ διαφορετικές εικόνες της δημοσιονομικής κατάστασης σε πολλά κράτη-μέλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλωστε και η έκθεση στο τέλος της αναφέρεται σε πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι χώρες θα μπορούσαν να δεσμευθούν για το ζήτημα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Θεωρώ ότι πολλά διαφορετικά πράγματα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν όμως εδώ πέρα προκειμένου να καταφέρουμε να βοηθήσουμε μονομένε χώρες και να αντιμετωπιστούν ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα δημοσιονομικά προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει. Και θα Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι οι αρνητικές οικονομικές εκτιμήσεις για το 2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με μια πολύ έντονη δύσκολη πολιτική κατάσταση σε ορισμένα κράτη-μέλη πολλές φορές οδηγούν σε χειρότερα αποτελέσματα σε οικονομική και κοινωνική πλευρά για πολλά κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, και όσον αφορά τα σχόλια τα οποία ήδη ακούσαμε από τους σκιώδεις, τον εισηγητή καθώς επίσης και άλλους συναδέλφους, νομίζω ότι όπως είπε και ο κύριος Παλώνε, η έκθεση αυτή μπορεί να βελτιωθεί. Υπάρχουν ε, πολλές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και που μπορούν τελικά να συμβάλλουν στο να βελτιωθεί η έκθεσή του. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε τροπολογίες οι οποίες προσπαθούν να τονίσουν όλα αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε πλέον στη διάθεσή μας όσον αφορά αυτή την αρνητική εξέλιξη των πραγμάτων συμπεριλαμβανομένου και του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν καταφέραμε να προβλέψουμε και να εφαρμόσουμε εκ των προτέρων δημοσιονομικές πολιτικές οι οποίες να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενσωματώσουμε στην έκθεση αυτή και κάποιες τροπολογίες οι οποίες ε, προσπαθούν να στείλουν ένα πολύ ηχηρό μήνυμα για την δύσκολη κατάσταση που βιώνουν πολλά και που θα συνεχίσουν να βιώνουν εφόσον εμένουμε απλώς σε μέτρα λιτότητας χωρίς να υπάρχει όμως ένα όραμα και ένα πρόγραμμα προκειμένου να επιστρέψουμε σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Και μια τελευταία παρατήρηση η οποία άλλωστε συνάδει και με τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα και τις ε, παρατηρήσεις που ήδη ακούσαμε, μολονότι έχουμε διαφορετικές πολιτικές απόψεις και κάνουμε διαφορετικές πολιτικές προτάσεις, θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους να λάβουν υπόψη τους τα όσα έχουμε στην πρώτη σελίδα της International Herald Tribune σήμερα. Αναφέρομαι δηλαδή σε ένα άρθρο με τίτλο ότι το κοινό χάνει πλέον την πίστη του, την, την εμπιστοσύνη του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχει κανένα ε, που να θέλει το λόγο. Θα επιστρέψω λοιπόν στον εισηγητή του κύριο Παλώνε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που έλαβαν το λόγο, διότι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή είναι ειδικά τη στιγμή να υπάρχουν ε, κοινέ απόψεις να συμμερίζονται οι τις απόψεις των ΔΕ. Γιατί τελικά όλοι μας επιθυμούμε να βελτιώσουμε μια κατάσταση η οποία εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στην Υπηρώμης. Δηλαδή υπάρχουν χώρες οι οποίες υποφέρουν εγώ λοιπόν είμαι υπέρ της ε, πολιτικής παροχής βοήθειας, και επίση υπέρ μια πολιτική η οποία αναμφίβολα πρέπει να οδηγήσει στην ανάπτυξη. Κοιτάξτε, ε, σαφώς και ε, πρέπει να είμαστε προσανατολισμένοι σε μια φορολογική πολιτική που κατευθύνεται προς την ανάπτυξη. Όμως δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Πρέπει να δούμε που θα περικόψουμε και πιο συγκεκριμένα θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοιες δημόσιες δομές σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη που είναι απαρχαιωμένες ε, και προκαλούν ανησυχία. Υπάρχει ε, πελατοκρατία, οικογενειοκρατία. Ξεκινάω από τη δική μου τη χώρα. Δεν θέλω να πω για άλλου. Άρα δηλαδή η δική μα η δουλειά, τουλάχιστον με τον δικό μου τον τρόπο σκέψης, η δική μας η δουλειά είναι να ε, ασχοληθούμε με την ανάπτυξη προσπαθώντας όμως παράλληλα στο βαθμό του δυνατού να μην επηρεάσουμε τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες γιατί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει τεράστιο βάρος στις επιχειρήσεις μεγάλο βάρος στα νοικοκυριά και αυτό αναγκαστικά οδηγεί στην ύφεση η κοινή αγορά στην Ευρώπη συρρυκνώνεται ακόμα και στη Γερμανία αν θέλετε ειδικά μάλιστα στο νότιο βόρειο τμήμα της Γερμανίας. Αυτές λοιπόν είναι σκέψεις που προφανώς και αναγκαστικά γίνονται. Άρα δηλαδή σύγκρουση υπάρχει ακόμα. Και θέλω να απαντήσω στο συνάδελφο Χέντελ. Ε, ίσως να μην εκφράστηκα εγώ καλά. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ένας που να λέει ή το άσπρο ή το μαύρο. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας μου. Ε, και με την έννοια ότι εγώ δεν εκφράζω συμφέροντα κανενός. Αν θέλετε, ε, από τη φύση μου είμαι λιγάκι πιο καχύποπτος, ίσως ε, να μην ελέγχθησαν καλά αυτά τα οποία είπα εγώ. Γιατί εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι εγώ δεν επιμένω άκαμπτα στο ξέρετε αυτό είναι και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ είμαι... Κάποιο ο οποίο επιθυμεί να διαπραγματεύεται, να συζητάει και όχι για να ε, χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και να επιμένει άκαμπτα στο να περάσει η δική του η θέση. Ε, προφανώς λοιπόν εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι να περάσει η θέση μου. Θα σας φέρω εδώ ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Μαζί με άλλους συναδέλφους υπάρχει η τροπολογία 69 σχετικά με τους φορολογικούς ε, πολλαπλασιαστές ε, δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές. Ε, Υπάρχουν θέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Τα πρέπει να είναι κάτω από το ένα αυτό ο περίφημο πολλαπλασιαστή. Αλλά α το συζητήσουμε. Δεν είναι δηλαδή ότι θα φτάσω στις συμβασικές προτάσεις λέγοντας ότι ξέρετε αυτή είναι η συγκεκριμένη γραμμή που πρέπει να επιβληθεί και κατόπιν τούτου δεν διαπραγματευόμεθα τίποτα. Δεν το λέω αυτό γιατί και οι περισσότερες ε, τροπολογίες που διάβασα επιθυμούν επιθυμώ εγώ τουλάχιστον να τη συμπεριλάβω στη σύνταξη τη τελική μου έκταση. Νομίζω ότι το ξεκαθάρισα αυτό με τον συνάδελφο κύριο Χέντελ. Του εξήγησα ότι εγώ δεν είναι ο χαρακτήρα μου ε, να κάνω κάτι τέτοιο. Και ξεκινώντας τον κύριο Χέντελ, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν. Στις 12 Νοεμβρίου θα ξανασυναντηθούμε. Ε, ελπίζω να κάνουμε καλή δουλειά και αν χρειαστεί θα υπάρξει και άλλη και μεθεπόμενη συνάντηση των ε, σκιωδών εισηγητών έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πλειοψηφία, να καταλήξουμε σε μια άποψη την οποία θα συμμερίζονται οι περισσότεροι συνάδελφοι και αυτό το λέω χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως προκατάληψη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ λέει και η Πρόεδρος. η ψηφοφορία θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου με στόχο να έρθουμε στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ Αλφρέδο. Και τώρα περνάμε στο σημείο 8 που είναι το πλαίσιο για την ανάκτηση είναι η έκθεση Γκίνερ Χόκμαρκ για την ανάκαμψη και την ανόρθωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Hockmark. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τους σκιώδεις συζητητέ. Είχαμε στο παρελθόν την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελα να αναφέρω σαν σημείο εκκίνησης. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύπλοκο θέμα, το πώς θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ένα πλαίσιο για τη διαχείριση των κρίσεων σε σχέση με τις τράπεζες. <clears throat> Είναι τεχνικό θέμα, είναι πολύπλοκο θέμα και μπορεί κανείς να είναι πολύ εύκολα ανοιχτός στην επίτευξη λύσεων, γιατί ακριβώς είναι τόσο πολλές οι απόψεις. Είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς όλα τα επιχειρήματα τα οποία διατυπώνται και να δει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους, αλλά το βασικό είναι να ξέρουμε ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος μας. Είπα προηγουμένως όταν συζητούσαμε το θέμα αυτό, ότι σε κάποιο βαθμό είναι ένα είδος ε, προσπάθειας ανάνυψης του καπιταλισμού, για να το πω με ομούς όρους, με την υποστήριξη της πολιτικής. Κανείς δεν μπορεί να διαμφισβητήσει ότι σε σχέση με τις τράπεζες πρέπει να εφαρμοστούν κανόνες που να μην οδηγούν μονάχα στην ιδιωτικοποίηση των κερδών, αλλά και την ανάληψη των ζημιών από τους ιδιοκτήτες των τραπεζών. Εδώ δεν πρόκειται για κάποιο σοσιαλιστή, χριστιανοδημοκράτη, φιλελεύθερο, ο οποίος θα διαφωνούσε με αυτή τη βασική άποψη. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την ανάγκη να έχουμε μια <clears throat> κοινή πολιτική αντιμετώπιση για τη φύση του προβλήματος. Και όλα αυτά μας οδηγούν σε μια διαδικασία με την οποία θα μπορέσουμε να αναζητήσουμε κοινέ λύσεις όταν συζητούμε στην Επιτροπή μας. Κάποια άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να επιτευχθούν σε σχέση με την σχεδίαση ενό πλαισίου για τη διαχείριση των κρίσεων είναι φυσικά το να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία όμως δεν δημιουργείται μονάχα από ένα πλαίσιο. Είναι απαραίτητο να υπογραμμίσω ότι στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο αντιμετωπίζουμε παράλληλα και άλλα θέματα συναφή που είναι πολύ σχετικά, όπως είναι το πλαίσιο CRD4 και το σχέδιο για την εγγύηση των καταθέσεων. Πρόκειται για τις, ε, τους λήθου λίθους στο λεγόμενο ενιαίο βιβλίο κανόνων που θέλουμε να θεσπίσουμε. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη να εξασφαλίσει ότι αυτός ο ενιαίος κατάλογος κανόνων θα μπορέσει να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα έφορο έδαφος αξιοπιστίας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε στη συνέχεια όλα τα θέματα τα οποία ουσιαστικά υποκρύπτονται πίσω από, το γενικό, από τη Γενική Επικεφαλίδα Τραπεζική Ένωση και είναι ακόμα πιο σημαντικά γιατί ο, το ενιαίο σύνολο κανόνων σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να διατηρήσουμε τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό της σε επίπεδο κανόνων. Έχω πει ορισμένε φορές στο παρελθόν κάπως ηρωνικά ότι όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα προσπαθούμε να επινοήσουμε μια νέα ένωση. Και στο τέλος θα φτιάξουμε μια ένωση η οποία είναι ένωση κατά του βήχα, κατά της γρήπης, κατά της πνευμονίας. Εμείς όμως χρειαστήκαμε να αγωνιστούμε σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο να έχουμε την τωρινή οικονομική ένωση και πολιτική ένωση στην Ευρώπη και είναι απαραίτητο να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό. Δεν θα πετύχουμε καλύτερη εποπτεία, μεγαλύτερη σταθερότητα με το να κατακαιρματίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένας αγρογωνιαίος λίθος της προσπάθειας μας να διατηρήσουμε τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να κάνουμε σοβαρές προσπάθειες για να ευδοκιμήσει αυτό το εγχείρημα. Μπορούμε όλοι να χαιρετήσουμε λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν. Είναι μια καλή πρόταση την οποία θα πρέπει να χαιρετήσουμε θετικά. Και θα θέλαμε όλοι να την είχαμε δει αυτή την πρόταση να έρχεται νωρίτερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ήρθε θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα ώστε να έχουμε αποτελέσματα στο θέμα αυτό μαζί με τα άλλα συναφή θέματα το ταχύτερο δυνατό και χωρίς να τα συνδέουμε κατά ανάγκη με όλα τα εκρεμή θέματα γιατί όταν προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα μαζί, προβλήματα μαζί για την Τραπεζική Ένωση και τις προσπάθειες της Ευρώπης στον τομέα αυτό, αν προσπαθούμε να τα λύσουμε όλα τα προβλήματα μαζί, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Είναι ήδη αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί η συμφωνία για το CRD4 και για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και αυτή η οδηγία επίσης θα έχει πολλές δυσκολίες. Άμα βάλουμε λοιπόν πολλά αυγά στο ίδιο καλάθι, τελικά μπορεί να καταλήξουμε να μην μπορέσουμε να επιτύχουμε την έγκριση όλων αυτών των μέτρων και να καταλήξουμε να υπονομεύουμε και τις προσπάθειές μας σε άλλους τομείς. Έχω τώρα κάποιε γενικέ κατευθύνσει στο σχέδιο έκθεση το οποίο παρουσιάζω στην Επιτροπή μα. Καταρχήν να εξασφαλίσουμε τη συνοχή και τη διατήρηση τη ενότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσει μια ρύθμιση που να καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, το οποίο είναι και το αντικείμενο και ο στόχο τη πρόταση Κομισιόν, είναι να διευκρινίσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε σωστά τις διαφορές οι οποίες μπορούν να προκύψουν μεταξύ των δράσεων των δημοσίων αρχών στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να αποφύγουμε το αρμπιτράζ το οποίο μπορεί να προκύψει, το κανονιστικό αρμπιτράζ το οποίο μπορεί να προκύψει από διαφορετικές ρυθμίσεις. Και επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν τελικά τράπεζες οι οποίες θα θεωρούνται πολύ μεγάλες για να ε, αποτύχουν, για να χρεοκοπήσουν. Θα θέλαμε να μην υπάρχουν αποτυχίες στον τραπεζικό τομέα, ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν πάντα δυνατότητες μια τράπεζα να βρεθεί σε κατάσταση αποτυχίας. Θα θέλαμε να έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει σε όλες τις τράπεζες να μπορούν να αποτύχουν ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε στη ζωή τον καπιταλισμό με τη βοήθεια των φιλελευθέρων, των σοσιαλιστών και των άλλων πολιτικών παρατάξεων. Αυτό θα σημαίνει επίσης ότι η ευθύνη για την δράση σε τέτοιε περιπτώσει μια τράπεζα η οποία αποτυγχάνει θα βρίσκεται στα χέρια των μετόχων των τραπεζών και όχι στις δημόσιες αρχές και μόνο. Όλα αυτά θα έχουν και ένα αποτρεπτικό χαρακτήρα θα επιτρέψει να αλλάξει και η φύση του τραπεζικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό εγώ έχω προσπαθήσει να διαχωρίσω διάφορες φάσεις σε ό,τι αφορά τις λύσεις ανάκτησης στο τραπεζικό σύστημα. Για μένα όσο μια τράπεζα εξακολουθεί να λειτουργεί είναι υπό την ευθύνη των συμμετόχων της και δεν πρέπει να υπάρχει μια φαιά περιοχή όπου παρεμβαίνουν οι δημόσιες αρχές και, δημιουργείται, και να δημιουργείται η εντύπωση στις αγορές ότι τα, οι κρατικές αρχές αναλαμβάνουν την ευθύνη. Γιατί πάλι αυτό θα δημιουργήσει σε προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια αποσαφήνιση της διάκρισης μεταξύ ανάκτησης και επίλυσης για τις τράπεζες. Ένα παράδειγμα είναι η ανάγκη να υπάρχει ένας ειδικό διαχειριστής μιας τράπεζας για μένα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβει η χώρα σε συνθήκε επίλυση μια τράπεζα. και σε αυτό το τμήμα τη νομοθεσία θα πρέπει να πάει. Ξέρω ότι αυτό συζητείται στο Συμβούλιο, αλλά από τη στιγμή που οι δημόσιε αρχέ παρεμβαίνουν σε μια τράπεζα, ο, η εντύπωση που δημιουργείται στι αγορέ είναι ότι αναλαμβάνουν το βάρο τη ευθύνη και οι δημόσιες αρχέ και ο φορολογούμενος. Γι' αυτό θέλω να έχω μια σαφή διάκριση μεταξύ της περιοχής ευθύνης των μετόχων και της περιοχής ευθύνης των δημοσίων αρχών. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα και το έχω αναφέρει και σε προηγούμενες συζητήσεις στην Επιτροπή μας, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει μια σαφής διαφορά του να υπάρχει μια τράπεζα η οποία αντιμετωπίζει κρίση και το να υπάρχει μια συνολική κρίση στο τραπεζικό σύστημα. Όταν μία τράπεζα βρίσκεται σε δυσκολία ή μία ή δύο τράπεζες είναι σε δύσκολες συνθήκες, αυτό είναι διαφορετικό από μία συνολική κρίση του συστήματος. Όταν έχουμε μία συστημική κρίση στο τραπεζικό σύστημα, αντιμετωπίζουμε συγχρόνως τεράστιες συνήθως μακροοικονομικές ανισομέρειες οι οποίες δημιουργούν απειλές για το συνολικό σύστημα. Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, μιας ύφεση, μιας κρίσης στις τιμές των, ε, των της ακίνητης περιουσίας κτλ. Είναι όλες αυτές τις περιπτώσεις όπου το πρόβλημα είναι εξωγενές, έρχεται από μια εξωτερική κατάσταση. Όταν μια τράπεζα όμως αντιμετωπίζει μια κρίση, είναι αποτέλεσμα των ενεργειών της των διοικητών και των μετόχων της τράπεζας που έχουν ε, κάνει λαθασμένες αποφάσεις, έχουν ακολουθήσει ένα λαθασμένο επιχειρηματικό μοντέλο. Είναι ένα εσωγενές λοιπόν πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η πρόταση της Κομισιόν είναι για μένα πολύ σωστή. Θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τέτοιες κρίσεις εσωγενείς, αλλά πρέπει να δούμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε και συστημικές κρίσεις. Η μορφή αυτών των συστημικών κρίσεων δεν θα είναι <clears throat> σταθερή, θα ήταν επικίνδυνο να πούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια συστημική κρίση με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Με τον τρόπο αυτό θα ξανακάνουμε το ίδιο σφάλμα που κάνουν πολλές φορές οι στρατιωτικοί όταν σχεδιάζουν με τα δεδομένα του προηγούμενου πολέμου. Γιατί η επόμενη κρίση δεν θα είναι σαν την τωρινή κρίση. Κάθε φορά η ιστορία αλλάζει. Και κάθε φορά η προηγούμενη κρίση μπορεί να αποτραπεί από την ε, νέα ρύθμιση και νομοθεσία, αλλά η επόμενη κρίση οφείλεται στα παραθυράκια τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν σε αυτή την νομοθεσία. Δεν νομίζω ότι κάποιος από μας μπορεί να πει ότι τέρμα δεν θα υπάρξει καμία χρηματοπιστωτική κρίση στο μέλλον. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε την σωστή και την πρέπουσα νομοθεσία για τα θέματα αυτά. Και γι' αυτό έρχομαι στις πρόσθετες προτάσεις μου, πέραν αυτών που πρότεινε η Κομισιόν. Προσπάθησα να διευκρινίσω ποια είναι η διαφορά μιας μεμονωμένης κρίσης σε μια τράπεζα και μιας συστημικής κρίσης και έχω παρουσιάσει προτάσεις για το πώς μπορούμε να καθορίσουμε τι ακριβώς είναι μια συστημική κρίση και πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τις παρεμβάσεις και τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες συστημικές κρίσεις. Πέραν των εργαλείων λοιπόν της Κομισιόν, η διαδικασία του bail-in, δηλαδή η ανάληψη ευθύνη από τους ίδιους τους ομολογιούχους και επίσης τα εργαλεία των δημοσίων αρχών οι ενέσεις κεφαλαίου, η μερική <clears throat> ιδιοκτησία από τις δημόσιες αρχές, ακόμα και η προσωρινή ανάληψη ιδιοκτησίας από τις δημόσιες αρχές. Θα ήθελα να πω προς την αριστερή πτέρυγα του, της Επιτροπής αυτής. Δεν είναι ότι ξαφνικά γίνομαι σοσιαλιστής. Απλώς θέλω να διευκρινίσω πότε θα είναι αποδεκτό να υπάρχει δημόσια παρέμβαση σε μια τράπεζα που αντιμετωπίζει δυσκολίες και πότε όχι. Γιατί όταν υπάρχει μια κρίση συνολική και όλη η οικονομία ενός κράτους μέλους ή μιας περιοχής βρίσκεται σε δυσκολία, είναι ε, σαφές ότι θα υπάρχουν εκκλήσεις για δημόσια παρέμβαση και πολλές φορές θα είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί ένα κλίμα φόβου και έλλειψης εμπιστοσύνης και ο μόνος τρόπος ανάκτησης της αξιοπιστίας να υπάρξει κάποια μορφή δημόσιας παρέμβασης. Αυτή είναι και η εμπειρία που είχαμε με συστημικές κρίσεις μέχρι στιγμής όσο είναι δυνατόν φυσικά πρέπει να αποφεύγουμε μια τέτοια δημόσια παρέμβαση. Όταν είναι απαραίτητο όμως τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι γίνεται η σωστή ε, παρέμβαση επί τη βάση μιας νομοθεσίας που αποτρέπει το να κάνουμε τέτοια πράγματα όταν δεν χρειάζονται, αλλά τα επιτρέπει όταν είναι απαραίτητα. Να ξέρουμε λοιπόν πότε μπορούμε να γίνουν δημόσιες παρεμβάσεις και πότε όχι. Και πολλές φορές πλανάται και μία παρεξήγηση ότι το να έχουμε μια νομοθεσία για δημόσια παρέμβαση σημαίνει ότι ανοίγουμε την πόρτα διάπλατα για δημόσια παρέμβαση. Εγώ όμω νομίζω ότι είναι καλύτερο να έχουμε μια νομοθεσία που θεσπίζει σαφή κριτήρια για το πότε πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση και πότε όχι <clears throat> και όταν είναι σαφέ τι ακριβώ θα σημάνει μια δημόσια παρέμβαση στον οικονομικό χώρο. Αυτή είναι λοιπόν μια από τι κατευθυντήριε αρχέ στην εκθεσή μου και θα ήθελα και ιδίω με του οικειώδει συζητητέ να έχω μια συζήτηση μαζί σα για το θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι η διαδικασία του bail-in, της ε, ανάληψης ενδεχομένων ζημιών από τους κατόχους ομολόγων. Τόνισα ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο πρέπει να έχουμε στο προστασιό μας. Αλλά το εργαλείο του bail-in είναι πάρα πολύ θετικό μέχρι τη στιγμή που θα χρειαστεί κανείς να το χρησιμοποιήσει. Έχει ένα αποτρεπτικό χαρακτήρα. Δεν προτρέπει στην ε, χρησιμοποίησή του, αλλά σε μια συστημική κρίση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα επιμόλυνσης και διάδοσης της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πιστεύω λοιπόν ότι και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουμε μια ευρεία συζήτηση, την έχουμε συζητήσει και με τους άλλους και συζητητές, πώς θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτό το εργαλείο για να του δώσουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία και επίσης να τον το έχουμε πιο πρόσφορο για χρησιμοποίηση σε συστημικές κρίσεις θα επανέλθω σε τεχνικό επίπεδο με τους σκιοδησίτες, αλλά πρέπει να κάνουμε και μια συζήτηση ευρύτερα στην Επιτροπή μας. Ενδεχομένω θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε σχέση με το επίπεδο, μάλλον με τα στοιχεία ε, χρέους των τραπεζών που μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι επιλέξιμα για τη διαδικασία του Μπέιλιν. Εγώ δεν ξέρω φυσικά ποια είναι η σωστή λύση στον τομέα αυτό. Ο Όλε Σμιτ με κοίταζε με πολλή απορία προηγουμένω. Αλλά είναι απαραίτητο να κρατήσουμε ένα ανοιχτό πνεύμα για το πώς θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τη διαδικασία του Μπέιλιν ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται με έναν τρόπο που είναι αξιόπιστος και αποτελεσματικός για την αντιμετώπιση κρίσεων και την επίλυση τραπεζών σε κρίση. <clears throat> Προσπαθώ να κλείσω λοιπόν την παρέμβασή μου κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι για τη χρηματοδότηση των, της επίλυσης των τραπεζών υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να <clears throat> είμαστε σαφείς ότι αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνεται να υπάρχει ένα ταμείο εκ των προτέρων εξάντε και όχι εκ των υστέρων. Αν υπάρχει επίλυση εκ των υστέρων, με χρηματοδότηση εκ των υστέρων, θα δείτε πολλές φορές ότι δεν έχουμε τα απαραίτητα χρήματα για να αντιμετωπίσουμε συστημικές κρίσεις. όταν βρεθούμε σε μια κρίση είναι πολύ δύσκολο να συλλέξει κανείς τα χρήματα που είναι απαραίτητα για την επίλυση των τραπεζών. Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο. Αν έχουμε χρηματοδότηση εκ των υστέρων, σημαίνει ότι οι τράπεζες οι οποίες τα έχουν καταφέρει καλά και έχουν αντέξει την κρίση, ουσιαστικά χρηματοδοτούν αυτές που τα έχουν κάνει θάλασσα και έχουν βουλιάξει. Βάζουμε τους καλούς να πληρώνουν για τους κακούς τελικά. ενώ θα έπρεπε να γίνεται ίσως το αντίθετο. Όλα αυτά είναι μια μορφή συλλογική ευθύνη που επιβάλλουμε στον τραπεζικό τομέα. Δεν αναφέρομαι σε κανένα συγκεκριμένα όταν το λέω αυτό. και προσπαθώ και πάλι να τονίσω στα πλαίσια της σοβαρότητας είναι απαραίτητο να υπάρχει μια χρηματοδότηση εξάντε για την επίλυση των τραπεζών που να έχει αξιόπιστο χαρακτήρα και να δημιουργεί γενικότερη εμπιστοσύνη. Αλλιώ δεν αξίζει τον κόπο καν να το συζητάμε το θέμα αυτό. Και τέλο, κυρία Πρόεδρε, για τα συστήματα <clears throat> εγγύηση καταθέσεων, εγώ έχω μια διαφορετική γραμμή από την Κομισιόν. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι εθελοντικό για τα κράτη-μέλη να μπορούν να δίνουν χρήματα σε άλλα κράτη τα οποία βρίσκονται σε δυσκολία. Φυσικά όμως αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και χαίρομαι και είμαι υπερήφανος που έχω την ευκαιρία να επομιστώ το θέμα αυτό. Είχα ήδη πολύ καλή εμπειρία στις ε, πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τους κοιόδες συζητητές. Περιμένω και τις αντιδράσεις τους τώρα, αλλά φυσικά και στην επερχόμενη συνάντηση μεταξύ σκιωδών εισηγητών και πιστεύω ότι αυτό το νομοθέτημα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Uh, σας ευχαριστούμε πολύ. Ποιος θα εκπροσωπήσει την ε, λύση η οποία απουσιάζει. Όνερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι η Ελίζα σας ζητά συγγνώμη που δεν είναι σε θέση να βρίσκεται εδώ πέρα. Θα πάρω και εγώ το λόγο λίγο αργότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ας δούμε τους άλλους και οδηγητέ τότε, πρωτού περάσουμε στους περαιτέρω μιλητές. Βόλφ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω στα γερμανικά γιατί έχουμε μία ομάδα επισκεπτών από την Αυστρία, συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο καθώς επίσης και διάφοροι διευθυντέ και επιχειρηματίες. Θα μιλήσω λοιπόν στα γερμανικά. Καλώ ήρθατε στι Βρυξέλλε. Όποιος λοιπόν ε, είχε αμφιβολίες ότι το θέμα αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα που συζητάμε σε αυτή τη θητεία, εχθές ε, θα άλλαξε γνώμη. Εχθές είχαμε τον ε, πρόεδρο τον, ε, του Γραφείου Διεθνών ε, Λογιστικών Προτύπων και εκείνος λοιπόν κατέστησε σαφές ότι είναι απόλυτα σαφές ότι πολλές τράπεζες αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Κομισιόν τώρα σχετικά αργά αλλά όχι πολύ αργά κατέθεσε επιτέλους αυτήν την πρόταση. Και εδώ συμφωνώ με τον προλαλήσαντα αυτά που είπε τα βρήκα ιδιαίτερα ισόρροπα και σκόπιμα. Και συμφωνώ με τον Γκούναρ ότι βεβαίως όλα αυτά χρήζουν και κάποιων βελτιώσεων. Δεν θα λοιπόν να φερθώ σε αυτά τα θέματα. Με αυτήν την πρόταση που κατατέθηκε, η πρόταση κατέθεσε και τη δική της την πρόταση για την Τραπεζική Ένωση. Η Τραπεζική Ένωση, η οποία αποτελείται από τρεις πυλώνες. Πρώτον, τον εποπτικό τομέα όπου θα έχουμε και ένα είδος ταμείου εκαθάρισης και αυτά τα οποία συζητάμε εδώ. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι να υλοποιηθεί οριστικά η Τραπεζική Ένωση αλλά να κάνουμε ε, τη συζήτηση για αυτά που μας έχει ήδη καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις όπου συμφωνώ με τον ε, Κουκμάρ και θα πω και κάποιες άλλες δικές μου απόψεις. Αυτό που είναι απόλυτα σαφές είναι ότι όλες οι τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καλύπτονται από αυτήν την οδηγία. Βέβαια πρέπει να διερωτηθούμε κατά πόσον στο πλαίσιο της επικουρικότητας τα ίδια τα κράτη-μέλη θα μπορούν να ορίζουν πόσο συχνά θα πρέπει να αναπτύσσονται τέτοια προγράμματα εξυγίανσης ή εκαθάρισης αν θέλετε. Καλό ε, αυτό που έκανε ο Χούκμαρ που εξαίρεσε κάποιους ε, θεσμούς και χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι λέει ότι τα συστήματα εξασφάλισης ε, των επενδύσεων παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και να πόκειται στα κράτη-μέλη να καθορίσουν κατά πόσον θα εμφανίζονται διασυνοριακά ως πιστωτές. Αυτό πρέπει να παραμείνει ως έχει. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω κάποιες παρατηρήσεις που θεωρώ ότι χρήζουν βελτίωσης. Η πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά αυτό το εργαλείο, το bailing it, αυτό το ε, στοιχείο διάσωσης με τα ίδια μέσα είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπε όμως και ο Γκούναρ, αυτή η ε, προληπτική επίδραση αυτή κάπως ε, θα χαθεί ε, όταν τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι αν τελικά ε, διαμορφώσουμε ένα τέτοιο εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα, το Belling in Instrument, θα βρούμε και τους κατάλληλους επενδυτές, γιατί οι άλλες τράπεζες προφανώς θα εξαφανιστούν. Δεν μπορούμε δηλαδή μια τράπεζα να την οδηγήσουμε, να την εξαναγκάσουμε να ε, συμμετέχει σε κεφάλαιο κινδύνου μιας άλλης τράπεζας. Γιατί με τον τρόπο αυτό ο κίνδυνος δεν εξαλείπεται, απλά μετακυλίεται. Και αυτό είναι λάθος. Πέρα από αυτό, δείτε και το εξή θέμα. Ποιος θα μπορούσε να είναι ένας δυνάμει επενδυτής. Παραδείγματο χάρη θα μπορούσε να είναι ασφαλιστικοί οργανισμοί. Γιατί οι ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν τους κινδύνους να τους ανακαλύψουν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αν κάτι δεν πάει καλά, τότε οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν κινδυνεύουν άμεσα. Παρόλα αυτά βέβαια οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να ε, διασφαλίσει ότι θα χειριστεί σωστά τα χρήματα των ασφαλισμένων. Μήπω θα έπρεπε να είναι συνταξιωτικά ταμεία. Μα δεν θέλουμε τα συνταξιωτικά ταμεία να συμμετέχουν σε αυτό το εργαλείο, το Μπέλινγκ και κάποια στιγμή να πει στου συνταξιούχου, ξέρετε, το χέτο χάσαμε τόσα χρήματα. Άρα δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούμε την εκείνη την μία μοναδική περίπτωση ποιος θα μπορούσε να είναι ένας καλός δυνάμει επενδυτής. Δεύτερον, τίθε το εξής ερώτημα. Ε, τα ε, τραπεζικά ομόλογα, τα οποία είναι μικρής διάρκειας, δηλαδή οριμάζουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Γκούμαρ λέει να εξαιρούνται αυτά που οριμάζουν σε έξι μήνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ επιφυλακτική και είπε μόνο ένα μήνα να εξαιρούνται αυτά του ενός μηνός. Εγώ νομίζω πάνω από ένα μήνα τώρα. Το κατά πόσον το 6 είναι σωστή, ο σωστό αριθμό, δεν είμαι σίγουρο, Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με τους εμπειρογνώμονε. Και τίθε και το εξή ερώτημα. Ε, ποια θα είναι η έκταση αυτού του εργαλείου του Bellingit. Μερικοί είπαν 5%. 5% και από το σύνολο των κεφαλαίων, όχι των κεφαλαίων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο. Αστάθμητα δηλαδή. Και αυτή νομίζω είναι η σωστή προσέγγιση. Ε, βέβαια το 5% έτσι αναφέρεται το στοιχείο, αλλά λένε να είναι πάνω από το 5%. Αν όμως λάβουμε υπόψη μας ότι στον κανονισμό περί δύο κεφαλαίων είμαστε πολύ αυστηροί και προσθέσουμε και αυτό το 5%, καταλαβαίνετε ότι φτάνουμε σε ένα τεράστιο ποσοστό. Ε, πολύ απαιτητικό. Πάρα πολύ απαιτητικό για ένα ε, κανονικό απλό χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο. Εγώ πιστεύω ότι τα ε, σχέδια διάσωσης και εκαθάρισης θα πρέπει να βασίζονται και σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Όχι μόνο όταν υπάρχει ενοποίηση, ε, όχι δηλαδή σε επίπεδο πολυεθνικής αλλά και σε επίπεδο θηγατρικής. γιατί αλλιώς ε, δημιουργείται ε, ένα πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται. Το επόμενο θέμα που εξετάζουμε είναι το εξής. Πού ακριβώς πρέπει να εγκατασταθεί αυτή η αρχή που θα επιλαμβάνεται εκαθαρίσεων. Στην εποπτεία θα πρέπει να είναι ένας ξεχωριστός φορέας μέσα στον έλεγχο αλλά κάπως οργανωτικά να έχει δική της αυτονομία και αυτοτέλεια. Αυτά είναι θέματα που χρήζουν ε, διευκρινήσεων. Συμφωνώ με τον Γκούναρ που λέει ότι εκτός από αυτό το εργαλείο το bail-in θα πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα παρέμβασης του κράτους. Νομίζω η ιστορία μόνη της έχει καταδείξει ότι είναι πολύ πιθανό τα επόμενα χρόνια, και δεν μιλάω τώρα για αύριο μεθαύριο, ας πούμε μετά από πέντε χρόνια να επανεμφανιστεί μια κρίση και τότε τα χρηματοπιστωτικά Ινστιτούτα δεν θα έχουν εξοπλιστεί ακόμα με τα απαραίτητα εργαλεία και ε, θα είμαστε και πάλι αναγκασμένοι να ζητήσουμε τη βοήθεια των φορολογουμένων και των κυβερνήσεων. Ε, υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που προτείνει ο Γκούναρ είναι λογικό, γιατί και εκείνο μιλά ε, από δική του εμπειρία. Στην Σουηδία κατά δεκαετία του 90 είχε σημαντική πολιτική θέση όταν τότε η Σουηδία αντιμετώπισε τη μεγάλη κρίση των τραπεζών και ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Το επόμενο θέμα και αυτό είναι σαφές. Αναφέρομαι στα ταμεία. Στόσο ε, στο ταμείο ε, των ε, εκαθαρίσεων όσο και στο επενδυτικό ταμείο των ε, και εκ των υστέρων μάλλον, εξάντε, εξάντε θα πρέπει να χρηματοδοτούνται, εκ των υστέρων με συγχωρείτε. Εδώ λοιπόν είναι σαφές ότι αυτό θα πρέπει να γίνει στα ίδια τα κράτη-μέλη. Μπορεί αυτό να αλλάξει μετά από 5-10 χρόνια. Όμως θα πρέπει να είναι ενιαίες οι ρυθμίσεις και το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι σε πολλά κράτη με τραπεζικέ εισφορές υπάρχουν σχέδια να συσταθούν αυτά τα ταμεία. Όμως χρησιμοποιούνται για διαφορετικού ε, λόγους. Στην Σουηδία α πούμε για να να ε, αποπληρωθεί το χρέος του κράτους, σε, άλλα, σε άλλες χώρες εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, όμως ε, το, η πρικοδότηση των ταμείων και οι απαιτήσει που θα ικανοποιούνται είναι διαφορετικές. Γι' αυτό οι κανόνες πρέπει να είναι ενιαίοι, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχουν ίση όροι ανταγωνισμού ανάμεσα στα χρηματοψηφιακά Ινστιτούτα και τις χώρες. Σε γενικές γραμμές, ο Γκούναρ καλά τα είπε, ε, είχε πολύ καλές συζητήσεις με τους σκιώδης ηγητές και είμαι σίγουρος ότι από κοινού θα καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική λύση. Ευχαριστώ. Um, I've Ευχαριστούμε πολύ ο Φιλίπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κούνερ, με εκνεύρισες γιατί είπες ότι υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία πως προς το ότι δεν θα, πρέπει οι, κοινων, οι πολίτες να πληρώνουν το τίμημα και δεν αναφέρθηκε καθόλου στην Ελλάδα. Ναι, αλλά το εννοούσα αυτό το πράγμα όμως. Ούτε αναφέρθηκα στην Ιρλανδία όμως. Λοιπόν, σοβαρεύομαι τώρα. Θα ήθελα να αφαιρθώ συγκεκριμένα στην έκθεσή σου, γιατί αναφερθήκαμε στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα ήθελα να επαναληφθώ. Όσον αφορά το εργαλείο το εργαλείο διάσωση με ίδια μέσα, συμφωνώ ότι το εργαλείο αυτό θα πρέπει να λειτουργεί στην πράξη. Δεν συμφωνώ όμω αν εσύ θέλει να το διαγράψει. Δεν νομίζω όμω ότι θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη μήνυα ακρόαση την οποία διοργανώσαμε. Ήταν μία από τι πιο επικοδομητικέ συζητήσει που είχα για το ζήτημα αυτό. Στα πλαίσια τη Επιτροπή ΕΚΟΝ, αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε είναι ένα εργαλείο bail-in, ένα εργαλείο διάσωση με ίδια μέσα, το οποίο να μπορεί πραγματικά να λειτουργεί. Και να μπορούμε λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε, να μπορούμε να αποφασίσουμε ποιο θα μπορεί να το χρησιμοποιεί, καθότι γνωρίζουμε ότι ε, το μεγαλύτερο εμπόδιο το οποίο έχουμε στη χρήση του είναι οι επιπτώσεις ε, ντόμινο. Το γεγονός δηλαδή ότι μπορεί ενδεχομένως κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιώντας το μέσο αυτό να μετακυλήσουν τα προβλήματα και την κρίση σε άλλα τέτοια ιδρύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε ποιοι θα μπορούν να το χρησιμοποιούν. Και αν πούμε ότι κάποια ιδρύματα δεν θα μπορούν να έχουν το bail-in, τότε δεν θα μπορούν να το χρησιμοποιούν ούτε σε πρωτογενές, ούτε σε δευτερογενές ή τριτογενές όμως επίπεδο. Αν δηλαδή χρησιμοποιούν κάποια μέσα παραγόγων. Αν λοιπόν μία τράπεζα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το εργαλείο τότε θα πρέπει να προβλέπεται μία γενική απαγόρευσή του σε οποιοδήποτε επίπεδο. Όσον αφορά τώρα τα μέσα παρέμβασης του κράτους, συμφωνώ μαζί σου ότι όντως αυτό είναι το τελευταίο σημείο στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε και κάτι θα πρέπει να πούμε και γι' αυτό. Δύο παρατηρήσεις εγώ έχω να κάνω. Πρώτον, για μένα ομοιάζει ουσιαστικά με μια κατάσταση μαζικής καταστροφής. Είναι σαν να έχουμε ένα πυρηνικό όπλο στα χέρια μας, το οποίο είναι καλύτερο να μην χρησιμοποιήσουμε, αλλά από την άλλη ο εχθρός ουσιαστικά θα πρέπει να γνωρίζει ότι ενδεχομένως μπορεί και να το χρησιμοποιήσεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να προβλέπεται μία αυτομα... αυτοματισμός όσον αφορά τη χρήση του εργαλείου αυτού. Δεύτερον, αυτό το οποίο πρέπει να μπορεί όμως να προβλέπετε είναι ότι είναι τελικά πυρηνικό όπλο, δηλαδή ότι ουσιαστικά θα εξαφανίσει εντελώς τους κατόχους ομολόγων. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες ήταν οι επιπτώσεις στους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτοχοι ομολογιών. Τρίτον, είδα ότι διέγραψες τις ε, διατάξεις αυτές οι οποίες λένε ότι αν το σχέδιο ανάκαμψης δεν ε, αντιστοιχεί, δεν συμφέρει την τράπεζα, τότε θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να επεξεργαστεί και η ίδια η τράπεζα ένα πρόγραμμα το οποίο ενδεχομένω να τη βοηθήσει να επιλύσει την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Έχουμε κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα, μάλλον δεν θα ήθελα να πούμε ότι έχουμε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τα οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί μια εξυγίανση, μια λύση. Περιόρισε λίγο το πεδίο εφαρμογή των τεστ αντοχή των τραπεζών. Προσπαθώντα να δημιουργήσει ένα ευρύτερο, μάλλον θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο να είχαμε ένα ευρύτερο επίπεδο τεστ αντοχή για τι τράπεζες και πιστεύω ότι ε, Υπάρχουν τρόποι προκειμένου οι τράπεζε να είναι λιγότερο εκτεθειμένες στον συστημικό κίνδυνο. Θα μπορούσαν οι τράπεζε να ήταν λιγότερο διασυνδεδεμένε. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να επηρεάσουμε το επίπεδο διασύνδεση το οποίο επιλέγει μια τράπεζα, ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Όσον αφορά τώρα την ε, αρχή εξυγίανση και τον επόπτη, θα ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο, θα διαρθρωθούν ως δύο διαφορετικοί παράγοντες, νομίζω το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ένα σύστημα αποτελεσματικό, το οποίο στην πράξη θα λειτουργεί και κάθε φορά που θέλουμε να ε, εξηγιένουμε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα, ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα, μια κεντρική αρχή που να μπορεί να πάρει σημαντικές εκτελεστικές αποφάσεις. Συμφωνώ ότι ε, μπορούμε να έχουμε σχέδια εξυγίανσης σε επίπεδο μήλου και σχέδια εξυγίανσης σε επίπεδο υποκαταστημάτων. Νομίζω πάντως ότι το Ταμείο Εξυγίανσης θα πρέπει να προχρηματοδοτείται, αυτό το έχουμε πει και στο παρελθόν, και θα αναφερθώ τώρα και στο ζήτημα της Τραπεζικής Ένωσης. Το να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό εποπτείας, έναν κοινό επόπτη για τις ευρωπαϊκές τράπεζες χωρίς να έχουμε προβλέψει ένα συγκεκριμένο σχέδιο ενιαίο επίλυσης και εγγύησης των καταθέσεων, τότε πραγματικά αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα σύστημα το οποίο δεν θα λειτουργήσει στην πράξη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή πρέπει να, παραμέν, να περιμένουμε όλο και περισσότερα νομοθετικά έγγραφα προκειμένου να ελοποιήσουμε αυτή τη βασική ιδέα. Νομίζω ότι με το κείμενο αυτό, με την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορούμε να υλοποιήσουμε το σύστημα αυτό, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει μόνο ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων ή ένα σύστημα εξυγίανσης, αλλά θα μπορέσει να λειτουργήσει και ως ε, σύστημα το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε οργανισμός επιθυμεί, προκειμένου να προβλέπεται ένα ενιαίο σύστημα επίλυσης. Αν δεν προβλεφθεί κάτι τέτοιο, νομίζω ότι το ίδιο το σύστημα δεν πρόκειται να λειτουργήσει στην πράξη. Και να ολοκληρώσω λέγοντας κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί λίγο πιο φιλοσοφικό. Είπες ε, ότι πολύ συχνά ως πολιτικοί Πρέπει να ακουγόμαστε πεπισμένοι για τον λέμε και που ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αισθάνεσαι πάρα πολύ σίγουρο και συμφωνώ μαζί σου και δεν θα πρέπει να λειτουργούμε σαν να ξέρουμε τα πάντα ή σαν να έχουμε στα χέρια μα μια απόλυτη επιστήμη. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν νομίζω όμω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δικαιολογία αυτή για να μην προχωρήσουμε σε πράξει το να λαμβάνει κανείς πολιτικές αποφάσεις ή επιχειρηματικές αποφάσεις προφανώς δεν είναι μια απόλυτη επιστήμη, δεν μπορεί να γίνει με έναν απόλυτο τρόπο. Το τι θα ενταχθεί στο νομοθέτημα αυτό ή όχι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενδεχομένως στην επιλογή αυτή να κάνουμε κάποια λάθη. Αλλά το να μην αλλάξουμε την υφιστάμενη αρτεκτονική είναι και αυτό μια επιλογή που θα έχει τις επιπτώσεις της. Αυτό το οποίο πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν είναι να δούμε τι θα συμβεί σε περίπτωση που δεν κάνουμε κάτι και κατά την άποψή μου αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί εναλλακτική επιλογή. Αλλάζοντα λοιπόν τις παραμέτρους του συστήματος, ενδεχομένως να κάνουμε κάποια σφάλματα και προφανώς θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι δεν έχουμε εμεί στα χέρια μας την απόλυτη αλήθεια και δεν γνωρίσουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει απολύτως το σύστημα. Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει ως δικαιολογία για την μη ανάληψη δράση η μη ανάληψη δράση, η έλλειψη κανονισμών μα έφεραν στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, την οποία δεν θέλουμε να ξαναδούμε στο μέλλον. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε σε δύο χρόνια πάλι μια συστημική κρίση. Πιστεύω λοιπόν ότι με την εργασία που θα κάνουμε στο κείμενο αυτό θα καταφέρουμε να αποφύγουμε τέτοιε κρίσει στο μέλλον. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, λέει και Πρόεδρος. Και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδους εργατε... Ε, εισηγητές για το έργο τους. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να σπάσουμε το φαύλο κύκλο που πρέπει να διασώζουμε τη μία τράπεζα μετά την άλλη. Εγώ συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Αλλά πρέπει να είναι σωστός ο... σωστό το σύνολο των κανόνων αυτών. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στον 20 πρώτο τριγωνικό διάλογο για τα θέματα αυτά και δεν νομίζω ότι η λύση είναι να παίρνει κανείς 150 σελίδες κειμένου το βράδυ στο γραμματοκιβώτιό του και να πρέπει να συζητήσει την επόμενη μέρα επί τη βάση αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε σωστά, αλλά χρειαζόμαστε και επαγγελματική αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα για τόσο σημαντικά θέματα. Εγώ συμφωνώ με τα ειδικά εργαλεία διαχείρισης ότι θα πρέπει να αφήνει την δίκηση των ε, τραπεζών στη θέση τους. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να τους αφήνουν στη θέση τους μέχρι να φτάσουμε ένα σημείο που δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν πια τα πράγματα και τότε περνάμε στο επίπεδο της επίλυσης του resolution. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια σχεδίαση η οποία να καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα. Εγώ ανησυχώ γιατί δίνεις στα κράτη-μέλη την εντύπωση να, που, να πούν ότι οι μικρότερες τράπεζες δεν, πρέπει να έχουν, δεν είναι υποχρεωμένες να έχουν κάποιο σχέδιο εάν πρέπει να περάσουν σε επίλυση. Αλλά είδαμε ότι πολλές φορές είναι μικρές τραπέζες οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν τις ιστομικές κρίσεις. Εντάξει, να έχουν ένα πιο ελαφρό καθεστώς οι μικρές τράπεζες, αλλά να πει ένα κράτος μέλος ότι ένα μεγάλο τμήμα του πιστοτικού τομέα δεν θα πρέπει να έχει σχέδια αντιμετώπισης κρίσης. Αυτό για μένα πηγαίνει πολύ μακριά. Συμφωνώ μαζί σου στο να υπάρχει και ένα είδος εξουσίας που αφορά μονάχα τις, ε, που αφορά τις εγκατεστημένες σε μια χώρα εταιρείε που να μπορεί δηλαδή ένα κράτο μέλο να αντιμετωπίζει αυτέ τι εταιρείε και όχι μονάχα αυτές οι οποίες προέρχονται από το ίδιο κράτο. Για το θέμα του Μπέιλιν, αυτό είναι τις διάσουμε ίδια μέσα, όπω λέγεται. Αυτό είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Στον τελευταίο διάλογο για, τις, για την κεφαλαιοχική επάρκεια, μας ε, είπε η Κομισιόν με διδακτικό τρόπο μη, μη ζητήσετε να έχουν ακόμα περισσότερο κεφάλαιο οι τράπεζες από ότι μπορεί κανείς να, περιμένει λόγω της φάσης του οικονομικού κύκλου. Αυτό είναι σίγουρα είναι υπερκυκλικό ε, ζήτημα. Όταν ζητάει κανείς σε μια εποχή δυσκολίας να έχουν περισσότερο κεφάλαιο οι τράπεζες, αυτό σίγουρα δεν βοηθάει. Εγώ βρίσκω ενδιαφέρουσα την ιδέα να υπάρχει μια χωριστή κατηγορία κεφαλαίου που είναι μονάχα ένα κεφάλαιο διάσωσης ώστε, με ίδια μέσα, ώστε, αν μια τράπεζα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει αυτό δεν θα οδηγήσει σε επιμόλυνση σε άλλες τράπεζες. Όλα αυτά είναι δελεαστικά. Αλλά το ερώτημα είναι ποιο συμμετέχει στο bail-in. Είναι τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια διάδοση Κάποιοι θα έχουν στα χέρια τους λοιπόν αυτό το εργαλείο. Αυτό θα έχει και οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις για να είμαστε πραγματικά ειλικρινείς. Αν ήμουνα ε, ασφαλιστική εταιρεία θα ήθελα να υπάρχει ένα είδος χρέος που μόνο εγώ να μπορώ να αγοράσω. Γιατί τότε θα ήταν περιορισμένες οι δυνατότητες άλλων να συμμετέχουν σε τέτοια κεφάλαια και θα είχε μια ειδική θέση η ασφαλιστική μετέρια. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να υπάρχει αυτό το ευάλωτο τμήμα του χρέους το οποίο να διακρατάται μονάχα από ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλα είδη πιστοτικών ιδρυμάτων. Πρέπει λοιπόν να, περιο... να κρατήσουμε το πλαίσιο του χρέους το οποίο μπορεί να υπόκειται σε μπέιλι να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο. Για μένα δεν είναι αποδεκτό να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει <clears throat> να πληρώνει μια τράπεζα, ε, να πληρώνει ο δημόσιος τομέα και οι καταναλωτές λεφτά για να σώσει μια τράπεζα όπως η Royal Bank of Scotland, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν ε, χρέο με μειωμένε εγγυήσει να μην βάζουν το χέρι στην ε, τσέπη τους. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε όλες τις τεχνικές πτυχές αυτού του θέματος και συμφωνώ μαζί σας ότι ορισμένε φορές Πρέπει φυσικά να υπάρξει δημόσια συμμετοχή στη διάσωση, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι μονάχα η τελευταία καταφυγή. Θα πρέπει να είναι μια τελευταία καταφυγή η οποία κερδίζει χρόνο και βοηθάει στη ρευστότητα, αλλά δεν οδηγεί σε μεταβίβαση της ιδιοκτησίας. Πολλές φορές οι τραπεζίτες είναι πολύ ανίκανοι στο να διχείζονται τις τράπεζες, αλλά η πολιτική μπορεί να είναι ακόμα χειρότερη για αυτά τα θέματα. Για το DGS τώρα. Κατανοώ ότι αν υπάρχει μία εκ των προτέρων χρηματοδότηση για το DGS, δηλαδή για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, ότι αυτό μπορεί να είναι θετικό. Αλλά όταν προσπαθούμε να έχουμε εναρμόνιση των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, κάνουμε αυτούς οι οποίοι είναι λιγότερο στεναροί, λιγότερο ισχυροί, να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με αυτούς που είναι πιο ισχυροί. Και οι χώρες όπου δεν υπάρχουν εθελοντικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων βρίσκονται σε χωριστή, σε τελείως διαφορετική κατάσταση. Ε, το σουηδικό μοντέλο, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να εξασφαλίσει ότι μια τράπεζα μπορεί να έχει ε, ένα απόθεμα εναντί του χρέου της. Αυτά λοιπόν δεν προστατεύουν όμως τους καταθέτες. Υπάρχει το θέμα της ε, προτίμησης που μπορεί να δοθεί εναντί των άλλων πιστωτών. Φαίνεται ότι σε άλλα μέρη της, του κόσμου οι καταθέτες, παραδείγματος χάρη στην Αυστραλία, έχουν προτίμηση έναντι των Ευρωπαίων καταθετών στην ίδια τράπεζα. Επομένως, οι εγχώροι καταθέτες τη χάνουν προστασίας με προτίμηση έναντι των ε, καταθετών που είναι από άλλα κράτη του κόσμου. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι ένα, ένας τρόπος θεμητού ανταγωνισμού και ίσης μεταχείρισης και θα πρέπει να βρούμε και κάποια λύση στα θέματα αυτά. Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο εδώ για τη δεσμευτική διαδικασία διαμεσολάβησης. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε ήδη στα πλαίσια της οδηγίας CRD. Αν δεν μπορέσει να ξεδιαλυνθεί το θέμα αυτό, όλα αυτά τα στοιχεία της Τραπεζικής Ένωσης, τα οποία είναι πολιτικά ευαίσθητα όπως τη διαμεσολάβηση, δεν θα ευδοκιμήσουν. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά για να τα διεκπαιρεώσουμε αυτά τα θέματα. Right. Uh, Πολύ ωραία, δεν έχω εδώ τον... Δεν υπάρχει κύριος Χουντής. Είναι εδώ ο κύριος Χουντής. Έχω λοιπόν τον κατάλογο των ομιλητών. Ε, να δω αν υπάρχει κανένας ε, άλλος. Θέλει κανείς άλλος να παρέμβει. Ξέρω ότι ε, θέλει να ε, παρέμβει η Κομισιόν, αλλά ε, μόνο αν υπάρχει χρόνος, γιατί η προτεραιότητα δίνεται καταρχήν στα μέλη. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Δυστυχώς είναι κλειστό το μικρόφωνο του ομιλητή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κούνα, ο οποίος ε, μας ε, παρουσίασε εκτενώς το όλο θέμα και γι' αυτό δεν θέλω να μπω εγώ σε λεπτομέρειες. Τα διάβασα όλα πολύ προσεκτικά και γίνεται λόγος για κρατική παρέμβαση αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα ε, για τα οποία ε, δεν συμφωνώ με τη θέση του Γκούνα. Παραδείγματος χάρη ε, στην αλληλένδεση μεταξύ κράτους και τραπεζών. Κυρίως σε περίοδους κρίσης νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο και έχουμε ζήσει αυτό το αρνητικό το οποίο προέκυψε στην Ισπανία, το καθοδικό σπιράλ. Γι' αυτό λοιπόν ε, αυτή τη ε, διασύνδεση τη βρίσκω πάρα πολύ προβληματική. Είπε προηγουμένως ότι θα πρέπει να έχουμε αυτό το εργαλείο, το bailing in, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συστημικούς ε, κινδύνους, ε, να υπάρχει αυτό το Ταμείο Επίλυσης, το Resolution Fund για τις ε, τράπεζες και κάθε χώρα να αναλαμβάνει μόνη της την ευθύνη για ένα θέμα. Εγώ πιστεύω ότι το κράτος πρέπει να διαδραματίζει ξεκάθαρο ρόλο. Πιστεύω λοιπόν ότι αν το όλο θέμα δεν είναι σαφές, αυτό είναι πρόβλημα. Ε, ίσως θα πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Βεβαίως ε, μπορεί κανείς να πει ότι ε, υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Ας δούμε λιγάκι την, ε, το αμερικανικό παράδειγμα. Βεβαίως δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με την Ευρώπη αλλά και στην Ευρώπη διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν προβλήματα σε ε, περιπτώσεις προβληματικών τραπεζών όπου τα προβλήματα μετακυλίστηκαν στο φορολογούμενο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποιος διαχωρισμός. Υπήρξαν 90 τράπεζες ε, που έπρεπε να στηριχθούν και αυτό προκάλεσε ε, μεγάλο κόστος ε, χρηματοδότησης στην Αμερική. Ίσως λοιπόν μπορούμε να μάθουμε μερικά πράγματα από τις δυσκολίες της Αμερικής. Η συζήτηση είναι πολύ περίπλοκη, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να καταβάλουμε προσπάθειες για να δούμε έτσι την εικόνα λίγο ευρύτερα. Αλλά κατά τα άλλα πρέπει να σας πω στηρίζω και εγώ αυτή την σοσιαλιστική άποψη ότι το κράτος πρέπει να διαδραματίσει ρόλο και γι' αυτό λοιπόν σε ευχαριστώ για αυτό που είπατε προηγουμένως. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πάρω το λόγο στη συνέχεια. Γκούνερ, η προσπάθειά σου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, κινείται στη σωστή κατεύθυνση και συμφωνώ με πολλά από τα όσα είπαν η Βίκη και ο Γόλφ. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του Μπέιλιν, του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, συμφωνώ με τις ανησυχίε που ακούστηκαν από του αδέλφου. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ε, θέλουμε να κάνουμε τους ασφαλιστικούς οργανισμούς εγγυητές τελικά για τις τράπεζες, όπως είπε και η Βίκη και στα πλαίσια της οδηγίας κεφαλαιακών απαιτήσεων νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το εργαλείο αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο κάθε φορά να λέμε ποιο ασφαλιστικό οργανισμός και για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να αναλάβει μια εγγύηση απέναντι σε μια τράπεζα. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να βρεθούν και ως προς το bail-in κάποιες εναλλακτικές μέθοδοι. Σε σχέση λοιπόν με τα όσα λέγονται στην τροπολογία 31, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους της τροπολογίας αυτής, θα πρέπει να καταβάλουμε πολύ σημαντικές προσπάθειες. Δεν είμαι πραγματικά πεπισμένη για το χαμηλό τίμημα το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί όπως λένε ορισμένοι στα πλαίσια του εργαλείου Μπέιλιν. Και όταν κάναμε την ακρόαση η γενική ιδέα ήταν ότι όντως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια κάποια ασφάλεια, αλλά αν πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω του εργαλείου αυτού η ίδια η τραπεζική κρίση, τότε πραγματικά το εργαλείο αυτό αντί να οδηγήσει σε εξυγίανση, ενδεχομένω να οδηγήσει σε μια μετάδοση, μετακύληση της κρίσης και σε άλλους οργανισμούς. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το 5% το οποίο προβλέπεται στο εργαλείο Bail-in. Συμφωνώ με τα όσα είπε ότι μια ενδεχόμενη επόμενη κρίση θα διαφέρει από την υφιστάμενη, επομένω οι διαδικασίε που θα πρέπει να προβλεφθούν θα πρέπει να είναι και αυτέ διαφορετικέ. Ωστόσο, νομίζω ότι θα πρέπει παρόλα αυτά να έχουμε συγκεκριμένε παγιωμένε διαδικασίε για συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία είμαστε ακόμα σε θέση να προβλέψουμε αρκεί να έχουμε την απαραίτητη ευελιξία για να προσαρμοστούμε και σε γεγονότα εκείνα τα οποία δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε. Για ποιο λόγο λοιπόν διέγραψε την σχετική διάταξη από, την, από το κείμενό σου, σε σχέση δηλαδή μετά όσο θα μπορούσε να κάνει η EBA, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Συμφωνώ επίσης με τις ανησυχίες τις οποίες εκφράζεις όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Αν δούμε την κατάσταση των μετόχων ή του κεφαλαίου, τότε να συμφωνώ ότι θα πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στο κεφάλαιο και όχι τόσο στη ρευστότητα. Ούτως ή άλλως η του κεφαλαιου τοτε συμφωνω οτι θα πρεπει να επιμεινουμε περισσοτερο στο κεφαλαιο και οχι τοσο στη ρευστοτητα ουτως η αλλως η ρευστοτητα υπάγεται στην οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα βρισκόμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση και ότι δεν θα επαναληφθούν τα όσα είδαμε στο παρελθόν και τα όσα είπε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων χθε, ότι βρεθήκαμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου οι τράπεζες δεν είχαν πλέον κεφάλαια. Καταλαβαίνετε ότι η έλλειψη κεφαλαίων οδηγεί αυτόματα σε κρίση ρευστότητας. Δεν νομίζω πάντως ότι ε, θα πρέπει να διαγράψουμε τα εργαλεία εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν ε, με την ε, ρευστότητα. Συμφωνώ πάντως ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το ζήτημα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Αν δούμε τα πράγματα, αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, Πάρα πολλοί στο παρελθόν λέγανε ότι η κρίση η οποία αντιμετωπίζουμε ήταν μια κρίση ρευστότητα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια κρίση ρευστότητα η οποία είχε προκληθεί από έλλειψη κεφαλαίων. Ο Πίτερ Σίμων έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση, πράγματι. Εγώ θα μιλήσω προσωπικά. Δεν έχουμε μια ενιαία θέση ακόμα με την Ελίζα Φερέ για τα θέματα αυτά. Θα σας πω κάποια προσωπικά μου σχόλια. Είναι πολύ θετικό το ότι στην έκθεση δεν υπάρχει κάποια μορφή ανάμειξης των διαφόρων ταμείων. Είναι χωριστό το θέμα της ε, της ε, προστασίας των ε, καταθετών και διαφορετικό το θέμα των ταμείων επίλυσης κτλ. Εδώ έχουμε βέβαια φαύλους κύκλους τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσουμε μεταξύ τραπεζικού χρέους και κρατικού χρέους. Πολλές φορές το κράτος πρέπει να σώσει τράπεζες οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλα προβλήματα, αλλά αυτό έχει αποτελέσματα και στο κρατικό χρέος. Επομένως τα τρία αυτά μέσα που αναφέρει ο Γκούναρ, το, η εγγύηση των καταθέσεων, η, ανάκτηση και η επίλυση στον τραπεζικό τομέα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού ώστε και η προστασία των καταθέσεων όπως και τα ταμεία επιλύσεως να έχουν αρκετή ε, χρηματοδότηση ώστε να περιορίσουν στο βαθμό του δυνατού την ανάγκη περαιτέρω κρατικής παρέμβασης. Και επίσης, επανέρχομαι στο εξής και πάλι. Αυτό το οποίο έχουμε ενώπιον μας αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι αυτά τα οποία μας προτείνει η Κομισιόν αυτή τη στιγμή θα έχουν το επαρκές επίπεδο για να καλύψουν αυτές τις ε, ανάγκες. Το 1,5 είναι, τα 100 είναι αυτό το οποίο προβλέπεται από την πρόταση της Κομισιόν. Ο Γκούναρ θεωρεί ότι πρέπει να φτάσει όμως το επίπεδο των ε, εγγυήσεων σε ένα σημείο που να μπορεί να καλύπτει και την ανάγκη της επίλυσης. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ υψηλότερες απαιτήσει για το Ταμείο, ε, για το ταμείο επίλυσης. Οι γερμανικέ τράπεζε έχουν ένα συνολικό επίπεδο καταθέσεων Μόνο, η, μόνο η Deutsche έχει ένα επίπεδο καταθέσεων 271 ε, δισεκατομμυρίων και το ταμείο το οποίο ε, θα μπορούσε να τα καλύψει αυτά βρίσκεται σε ένα επίπεδο μονάχα 78 δισεκατομμυρίων για να μπορέσει κανείς να λάβει υπόψη και άλλες ε, τράπεζες, να έχουμε ένα ταμείο το οποίο φτάνει συνολικά μόνο στα 69 ή 70 δισεκατομμύρια, αυτό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ε, ασφάλισης καταθέσεων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ακόμα και οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, κατά τη δική μου άποψη, δεν είναι επαρκείς για να μπορέσουν να καλύψουν τα θέματα αυτά. Εμείς για το Ταμείο της Επίλυσης θέλουμε να αποφύγουμε τη χρήση αυτού του συστήματος και να υπάρχει δυνατότητα με ίδια μέσα οι τράπεζες να επιλύουν τις συνθήκες αυτές. Όλα. Όλα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα μιλήσω τη δική μου γλώσσα αυτή τη φορά, γιατί πιστεύω ότι όταν είναι Σουηδό ο εισηγητή, μπορούμε επιτέλου να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γλώσσα. Βάλτε τα ακουστικά σα λοιπόν. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή, να ευχαριστήσω τον Κούναρ για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ καλή έκθεση. Νομίζω ότι έχετε εστιάσει σε ένα αριθμό δύσκολων θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και επίσης καταγράφεται και το γεγονός ότι υπάρχουν και φαιές περιοχές και υπάρχουν προβλήματα. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Και επίσης χαίρομαι που είναι μετριοπαθή τη προσέγγιση σας και σα υποστηρίζω. Και ο συνάδελφός μου ο οποίο ε, μίλησε για το θέμα αυτό, ίσως δεν πιάσατε το αστείο που είχε να κάνει με την εσωτερική πολιτική ζωή της Σουηδίας. Αλλά αυτά είναι δικά μας θέματα, είναι η εσωτερική μας κουζίνα. Πριν από δύο εβδομάδε, έλαβε χώρα εδώ πέρα μια πολύ καλή ακρόαση και ο Μπολτ Λούντγκρεν ήταν ο αρμόδιος υπουργός της Σουηδίας στη δεκαετία του 1990 όταν ο Γκούναρ και εγώ ήμασταν βουλευτές στο Σουηδικό Κοινοβούλιο δεν ήταν μια πολύ εύκολη εποχή και ο Λούντγκρεν ήταν αυτός ο οποίος διατύπωσε τότε αυτές τις προτάσεις και αντιμετώπισε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στη χώρα μας τότε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Η τράπεζα Μπέλεμπεργκ στην Σουηδία, που ήταν μια από τις πιο σημαντικές στην Σουηδία αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα. Ουσιαστικά είχαν πάει στο Υπουργείο οι επικεφαλής της τράπεζας, φοβόντουσαν θα καταρρεύσει η τράπεζά του και χάρη στον Λούντγκρεν, τον Μπολούντγκρεν, μπόρεσε να υπάρξει μια λύση στο πρόβλημα αυτό και το είχε τονίσει στο παρελθόν τότε στην ακρόαση ότι πολλές φορές πήγε στο Σουηδικό Γραφείο για τα θέματα χρέους και τους είπε ποτέ μα ποτέ μα ποτέ δεν ε, πρέπει να πείτε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τα δημόσια κονδύλια για να αντιμετωπιστεί αυτή μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό έλεγε ο Γκούνερ προηγουμένω και όλε κάπω ηρωνικά συμφώνησε μαζί του. Αυτό μου δείχνει εμένα ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και γιατί τέτοιου είδου σενάρια, γιατί τέτοιε καταστάσει μπορούν να προκύψουν. Και βλέπω τώρα την τροπολογία παραδείγματο χάρη 40 στο εγγραφό σου Γκούνερ που μιλάει για το συστημικό κίνδυνο. Πιστεύω ότι εδώ βρίσκεται μια φαιά περιοχή, βρισκόμαστε σε μια φαιά περιοχή. Και πολλοί συνάδελφοι το είπαν αυτό. Πώς θα μπορούσες να αξιολογήσεις τις ανάγκες εκεί, πότε ακριβώς ισχύει μια συστημική κρίση και πότε όχι. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε ίσως στο μέλλον. Είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει κανείς όχι μονάχα τεχνικά αλλά και πολιτικά σε κάποια λύση. Γιατί από πολιτική άποψη είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό. Και κάτι ακόμα, Γκούνερ. Πότε θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει ένας κίνδυνος διάδοσης μιας κρίσης, μιας δυσκολίας. Γιατί αυτό είναι το επίμαχο θέμα στις συστημικές κρίσεις. Ξέρω ότι οι Πολιτείες το αντιμετώπισαν αυτό το θέμα με διαφορετικό τρόπο. Στρέφομαι προς τον Έλλο Λούντιξον. Είναι ομοσπονδιακό κράτος οι Πολιτείες και έχουν διαφορετικές μεθόδους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν κατακλείδη, να σας πω το εξή. Εγώ ήμουνα στο παρελθόν αρμόδιος για την οδηγία για την αποζημίωση των επενδυτών και εξακολουθώ σε κάποιο βαθμό να παρακολουθώ το θέμα αυτό, το οποίο όμως τώρα έχει περάσει τον κύριο Σέμον για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχουν μέτρα εξάντε εκ των προτέρων. Αναρωτιέμαι όμως το εξή. Μιλήσατε για εθνικά συστήματα Είπατε ότι πρέπει να υπάρχουν εθνικά συστήματα, εγχώρια συστήματα τα οποία θα διατηρηθούν και δεν θα πρέπει να θέσουμε αυτά τα συστήματα ένα βιβόλο και δεν πρέπει να θέσετε σε κίνδυνο και τους φορολογουμένους για να σώσει μια χώρα, μια άλλη χώρα πραγματικά. Αναρωτιέμαι όμως σε κάποιες καταστάσεις όταν όλα τα πράγματα βρίσκονται σε αβεβαιότητα, όταν υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στον οικονομικό τομέα Μήπως θα πρέπει κάποτε να χρησιμοποιείται και η έννοια τη αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με το Ταμείο Αποζημίωσης των Επενδυτών, να υπάρχει μια χρηματοδότηση εκ των προτέρων, ώστε εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να υπάρχει η υποχρέωση να βοηθήσετε μια άλλη χώρα εάν είναι απαραίτητο. Όχι κατά ανάγκη το 10% το οποίο προβλεπόταν αρχικά, αλλά 5%. Εδώ είναι το ερώτημα λοιπόν το οποίο θέλω να σου θέσω, Γκούνερ, Σε ρωτώ δεν θεωρείς ότι χρειάζεται να υπάρξει και ένας μηχανισμός αλληλεγγύης και για αυτό το σενάριο. Και να σου υπενθυμίσω ότι υπάρχει σήμερα στις σουηδικές εφημερίδες ένα άρθρο για τον George Soros, ο οποίος επιχειρηματολογεί <clears throat> ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επανέλθει επιτέλους, λέει, στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τέσσερις δύσκολες εποχές να υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν μπορούμε να καθόμαστε ο καθένας στη δική του χώρα με τι δικές τους δυνατότητε και εργαλεία. Η Σουηδία τα καταφέρει καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να συμμετέχουμε στο να βοηθήσουμε τους άλλους αυτούς οι οποίοι ήταν οι Να τους πούμε ότι έφταξαν, ότι έκαναν λάθος, αλλά αν δεν καταλαβαίνουν ότι αυτοί έφταξαν, αν έχουν εμπλακεί και αυτοί σε μια αρνητική σπήρα προς τα κάτω. Εκεί ίσως χρειάζεται αλληλεγγύη να βοηθήσουμε και τους άλλους για να μπορούμε όλοι να βγούμε από τη δύσκολη κατάσταση, από τη λούμπα στην οποία βρισκόμαστε. Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Μήπως πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστούμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να πάρει το λόγο εφόσον επιθυμεί Μάριο. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο. Όπως και πολλοί ομιλητές θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γκούναρ για την έκθεση αυτή, για την εργασία την οποία έχει κάνει. Είχαμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε κι άλλες στο μέλλον και ξέρετε ότι συνηθίζουμε εμείς να συνεργαζόμαστε εκ του σύνεγγις με τους εισηγητές για τα ζητήματα αυτά. Συμφωνώ με τον κύριο Βολφ Κλίντς που είπε ότι το ζήτημα αυτό είναι από τα πιο σημαντικά, όντως είναι. και ουσιαστικά συντοποιεί κανείς, ε, όπως πολλές φορές σε συστήματα σωληνώσεων, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το σύστημα αυτό όταν μόνο όταν δεν λειτουργεί. Σε περίπτωση λοιπόν οικονομικής κρίσης συνειδητοποιούμε ότι χρειαζόμαστε απαραίτητα ένα τέτοιο σύστημα. Πρέπει λοιπόν να το πετύχουμε απολύτως. Δύο πράγματα θέλω να πω ιδιαίτερα θετικά. Καταρχάς, Συμφωνώ ιδιαίτερα με την έμφαση που τόσο συγητή όσο και οι συναδελφοί του δίνουν για την εκ των προτέρων χρηματοδότηση. Συμφωνούμε απολύτω με την προσέγγιση αυτή. Και η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω έχει να κάνει με το ότι πράγμα το οποίο είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένω να καθυστέρησε να υποβάλει την πρόταση αυτή για μερικού μήνε. Πιστεύω πάντως ότι πρέπει αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή η πρόταση έχει υποβληθεί, να αρχίζουμε να εργαζόμαστε γρήγορα. Να σας πω λοιπόν και τη δική μας την άποψη. Σε ποιους τομείς θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Πρόκειται για τομείς ε, στους οποίους αναφέρεται προφανώς η έκθεση και είμαι πεπισμένο ότι θα συνεχιστεί επικοδομητικά η συζήτησή μας. Να σας πω τώρα για ποιο λόγο θεωρούμε ότι κάποιοι τομείς είναι ιδιαίτερα ε, σημαντικοί. Ο πρώτος και πιο σημαντικός είναι ο τομέας αυτός που έχει να κάνει με τις απαιτήσει όσον αφορά την επίλυση, την ανάκαμψη, την εξυγίανση των τραπεζών. Πιστεύω ότι οι απαιτήσει όσον αφορά την ανάκαμψη και την εξυγίανση, τα σχέδια ανάκαμψη και εξυγίανση δεν θα πρέπει να υποβαθμιστούν και πιστεύω ότι όλη η προληπτική δράση που μπορεί να υπάρχει, όλες οι προληπτικές αρμοδιότητες θα πρέπει να συνεχίσουν να παραμένουν στο κείμενο. Όταν παρουσιάσαμε την πρόταση αυτή είχαμε πει ότι η συγκεκριμένη πρόταση απαρτίζεται από τρεις τομείς. Σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης, πρόορη δράση και χρηματοδότηση, καθώς επίσης και το εργαλείο Bailin, το εργαλείο διάσωσης μίδια μέσα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στον ε, ειδικό αυτό διαχειριστή μάνατζερ, ο οποίος προβλέπεται και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο οποίος θα μπορούσε να παρέμβει ακόμα και στην ε, φάση της πρόορης ε, παρέμβασης γιατί ακριβώ έχουμε δει ότι υπάρχουν ορισμένε χώρε που ήδη έχουν θεσμοθετήσει ένα τέτοιο σύστημα και το οποίο λειτουργεί ικανοποιητικά. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να παραμείνει το σύστημα αυτό. Λοιπόν, σε ποια άλλα σημεία θα πρέπει να επιμείνουμε. Όταν αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία διασυ... ε... διάσωσης, εξυγίανσης μάλλον, σαφώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο bail-in. Είναι πολύ σημαντικό το εργαλείο αυτό να λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο κύριο Χόκμαρκ είπε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά θα πρέπει το εργαλείο αυτό να λειτουργεί τη στιγμή που θα το χρειαστούμε. Εκεί έγκυται πραγματικά η δυσκολία και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογή όσον αφορά το bail-in. Φαντάζομαι ότι θα γίνει μια συζήτηση σε σχέση με το πεδίο εφαρμογή. Εμεί θεωρούμε ότι το ευρύτερο πεδίο εφαρμογή εγγυάται τη σωστή λειτουργία του συστήματο αυτού όταν ακριβώ απαιτείται η χρήση του. Δεύτερον, επέκταση του συνόλου εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο κύριος Χόκμαρκ αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό με τρόπο πολύ συγκεκριμένο. Θα ήθελα και εγώ να είμαι ιδιαίτερα σαφής. Είμαστε σαφώς υπέρ αυτού του toolbox, αυτού του συνδυασμού εργαλείων, αρκεί να είναι σωστά πλαισιωμένος. Τι εννοώ λέγοντα σωστά πλαισιωμένος τασόμαστε υπέρ των εργαλείων αυτών γιατί ουσιαστικά δίνουν μια κάποια νομική βεβαιότητα. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά όμω, θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένους κανόνες. Είναι πολύ καλύτερο να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία αυτά όταν διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί δίνουν μια μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα. Θα πρέπει όμως να έχουμε και κάποιες διασφαλίσεις. Πρώτον, ότι τα εργαλεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε έσχατες περιπτώσεις, αφού δηλαδή έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες εναλλακτικέ. Και δεύτερον, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αυτά, δεν θα αυξηθεί ιδιαίτερα το χρέος το οποίο προέρχεται από την δημόσια χρηματοδότηση. Ξέρετε ότι ε, επεξεργαζόμενοι την πρόταση αυτή, θέλαμε ουσιαστικά να προσέξουμε ιδιαίτερα τη διασύνδεση η οποία μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο δημόσιο χρέος και τις τράπεζες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και επεξεργαζόμενοι τώρα το κείμενο αυτό να εξασφαλίσουμε σωστή ισορροπία στη διασύνδεση αυτή. Αναφερόμενος τώρα στην ίδια την έκθεση, βλέπω ότι στην αιτιολογική σκέψη, στεκτιμώντας, γίνεται μία προσπάθεια να αποσαφινιστούν όλα αυτά τα σημεία. Ενδεχομένως όμως και το διατακτικό θα μπορούσε να αποσαφανιστεί λίγο περισσότερο και να συνάδει περισσότερο με τεκτιμώντας. Μία ακόμα παρατήρηση που θέλω να κάνω, νομίζω ότι ο Φίλιπ Λαμπέρτ αναφέρθηκε σε αυτό. Το status quo. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση από την οποία θέλουμε να ξεφύγουμε η υφιστάμενη κατάσταση, η τρέχουσα κατάσταση είναι μια κατάσταση με ένα περιορισμένο νομοθετικό πλαίσιο. Έχουμε κρατική παρέμβαση απουσίας, απουσία κανόνων. Θέλουμε να ξεφύγουμε πλέον από την αβέβαιη αυτή κατάσταση και νομίζω ότι μέσω της πρότασης αυτής μπορούμε να ξεφύγουμε. Ας μην ξεχνάμε και σε σχέση με το G20 αυτής, αφού του Σαββατοκύριακου ότι υπάρχουν σαφώς κάποια εργαλεία τα οποία απορρέουν από κανόνες που έχει προβλέψει το G20. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και στον τομέα αυτό όπως και σε άλλους τομείς να καταλήξουμε σε κανόνες οι οποίοι θα συνάδουν με πράγματα τα οποία έχουν αποφασιστεί σε επίπεδο G20 κατακλείδη να ευχαριστήσω τον εισηγητή καθώς επίσης και όλους τους σκιώδεις εισηγητές και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία μαζί σας που θα οδηγήσει προφανώς σε ένα ιδιαίτερα ποιοτικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, um, and, um, thanks. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Γκούνερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις που γίνανε από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ο Φιλίπ έχει φύγει. Θα ήθελα απλώ να του πω ότι θα ήθελα όλοι οι πράσινοι ή οποιοδήποτε άλλοι εκπρόσωποι πολιτικών ομάδων να συνταχθούν με την προσπάθεια την οποία κάνω στην ε, έκθεση αυτή. Υπάρχουν κάποιοι κοινοί παρανομαστές που νομίζω ότι ε, μπορούν να εφαρμοστούν από όλου. Να συμφωνήσω απόλυτα μετά όσα μόλις τώρα μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νομική βεβαιότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Για δύο λόγους. Η νομική βεβαιότητα σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε δράση όταν αυτό απαιτείται, χωρίς ε, ουσιαστικά να αφισβητεί τη δράση σας και νομική βεβαιότητα σημαίνει επίσης ότι έχετε και την ευελιξία να αναλάβετε δράση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι μελλοντικέ κρίσεις θα είναι διαφορετικές ή η κρίση διαφέρει από τη μία περιοχή στην άλλη. Θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπε ο κύριος Λούντβικ δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε εσωκομματικές καταστάσεις της Σουηδίας. Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι συνάδει η στάση του με τις δικές μου αποφάσεις όσον αφορά την επέμβαση του κρατικού τομέα στις τράπεζες. Ουδέποτε ουσιαστικά έχω ακούσει έναν σου Σουηδό να μιλάει τόσο καλά για τις Αμερικανικές τράπεζες όσο σήμερα και αναφερθώ συγκεκριμένα παραδείγματα όσον αφορά τον Αμερικανικό τραπεζικό τομέα. Οι Lehman Brothers δεν βρισκόταν προφανώς στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αν είχαμε αποφύγει την ε, περίπτωση της Lehman Brothers, αν την είχαμε προβλέψει, θα είχαμε καταλήξει σε μια νομοθεσία πολύ καλύτερη και μια νομοθεσία η οποία θα επέτρεπε μια πολύ πιο αποτελεσματική επέμβαση του δημοσίου τομέα. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα είχαμε γλιτώσει τεράστια ποσά χρημάτων. Θα είχαμε αποφύγει αυτό το μέγεθος της κρίσης. Θα είχαμε καταφέρει να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε καλύτερα το αμερικανικό σύστημα, να δούμε τι θετικά στοιχεία μπορούμε να αποκομίσουμε, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι τελικά η κρίση ξεκίνησε μετά όσα συνέβησαν στην Lehman Brothers και ουσιαστικά ξεκίνησε από όλου αυτού οι οποίοι θεωρούσαν ότι ε, η τράπεζα αυτή δεν θα κατέρε και τελικά την άφησαν να καταρρεύσει. Τα συστημικά προβλήματα τα οποία ξεκίνησαν από την κατάρρευση αυτή ήταν καταστρεφτικά μετά και την πραγματική οικονομία. Α είμαι όμω σαφή, δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να δημιουργήσω ένα σύστημα το οποίο δεν υφίσταται, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι στα πλαίσια μιας κρίσης σαφώς θα υπάρχουν αιτήματα δημόσιας επέμβασης και δημόσιας χρηματοδότησης. Άκουσα τις παρατηρήσεις που κάνανε οι συναδελφοί μου. Και ξέρουμε πώς ήταν τα πράγματα σε καλύτερες εποχές, κάθε φορά που υπήρχαν κρίσει. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούσε το σύστημα τότε. Αν όμως να ακολουθήσουμε του παλιού παραδοσιακού κανόνε, τότε ουσιαστικά οδηγούμε τι τράπεζε στην καταστροφή. Και νομίζω ότι την εποχή που συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούσαν πραγματικά να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο που θα είχε μια και κατάρρευση τραπεζών στην ε, γενικότερη οικονομική κατάσταση. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τα ζητήματα αυτά και να κάνουμε τη σχετική συζήτηση. Κάθε φορά που βλέπουμε ότι πρέπει να αναλυφθεί δράση, η δράση αυτή θα πρέπει να διέπεται από κανόνες είναι πολύ καλύτερα να διέπεται από συγκεκριμένα κριτήρια. Ο οι Σμιτ με ρώτησε ποια είναι τα κριτήρια αυτά. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος ορισμός αυτή τη στιγμή για το τι είναι συστημικός κίνδυνος και συστημική κρίση. Έχουμε λαμπρούς οικονομολόγους οι οποίοι έχουν συμβάλει πάρα πολύ στους ορισμούς αυτούς. Θα μπορούσαν όμως να βελτιωθούν. Και βλέπω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πιο ικανοποιημένη με το μεταεκτιμώντας με την αιτιολογική σκέψη της έκθεσης αυτής και όχι τόσο με διτακτικό. Ενδεχομένω θα πρέπει πραγματικά να επικεντρωθούμε σε κάποιους ερωισμούς που έχουμε ακριβώς στο τμήμα αυτό της έκθεσης. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να εντάξουμε την δημόσια επέμβαση ως ένα εργαλείο που θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε, αλλά θα πρέπει αυτή η επέμβαση του κράτους να διέπεται από συγκεκριμένα κριτήρια και συγκεκριμένους κανόνες. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα το εργαλείο Bailin, το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα. Ο, ο, ο Φιλίπ αναφέρθηκε στον αποτρεπτικό χαρακτήρα που μπορεί να έχει το εργαλείο αυτό. Είπε ότι ομοιάζει με πυρηνικό όπλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως κάθε φορά που βρισκόμαστε σε μία βαθιά συστημική οικονομική κρίση να μην έχουμε μόνο μία εναλλακτική για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή. Ακόμα και αν έχουμε το εργαλείο θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Αν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις, τότε τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρώ λοιπόν ότι το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα, το εργαλείο είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο διάσωσης που πραγματικά θα αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα όσον αφορά την τραπεζική κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσει να χρησιμοποιείται. Θεωρώ ότι ε, θα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα αποβεί αξιόπιστο ακόμα και σε πολύ δύσκολες οικονομικές στιγμές. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ και για την ακρόαση που είχαμε, αλλά και για τη συνάντηση των ιστών όπου μιλήσαμε συγκεκριμένα για το εργαλείο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα εργαλείο, αλλά το εργαλείο αυτό θα πρέπει να είναι αξιόπιστο. Αυτό ακριβώς πρέπει να εξασφαλίσουμε. Πολλές αναφορές γίνανε για διάφορα σημεία της έκθεσης και ιδίως όσον αφορά τους κανόνες ρευστότητας. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι πάλι και εδώ πέρα να έχουμε μία νομική βεβαιότητα και να καταφέρουμε να ευθυγραμμίσουμε τους κανόνες ρευστότητας μετά όσα προβλέπονται στην Οδηγία για τις Κεφαλαϊκές Απαιτήσει Υπαριθμών 4. Ξέρετε όμως ότι άλλο ρευστότητα και άλλο φεργιότητα. Ο Φιλίπ νομίζω ότι ε, αναφέρθηκε στο ότι ε, τα σχέδια ανάκαμψης μπορούν να τροποποιηθούν ε, με βάση το ποια αρχή επίλυσης ή εξυγίανσης προχωράει στα προγράμματα αυτά. Νομίζω ότι τα πράγματα διαφοροποιούνται. Αν οι δημόσιες αρχές είναι αυτές οι οποίες επεμβαίνουν στις τράπεζες και τις καλούν υιοθετήσουν μια στρατηγική για τις επενδύσεις τους, τότε μπορεί να λειτουργήσει θεωρητικά καλά το σύστημα αυτό, αλλά Τι συμβαίνει στην πράξη όταν ε, η αρχή εξυγίανση δεν δίνει τελικά καλές συμβουλές, αν τελικά δεν βοηθά στην πράξη, αν τελικά της δημιουργεί άλλα προβλήματα. Η Βίκη είπε ότι ε, χειρότερα από τους τραπεζικούς στην διαχείριση των τραπεζών είναι η ίδια πολιτική και ότι ενδεχομένω ε, θα πρέπει να αφήσουμε άλλου ανθρώπου εκτό τραπεζικού τομέα να ασχοληθούν με το τομέα αυτό, μπορεί να γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα. Α μην συγχαίουμε όμω τι διαφορετικέ αρμοδιότητε. Όσο οι τράπεζε βρίσκονται υπό την ευθύνη των μετόχων τους, τότε θα πρέπει να σεβαστούμε το σύστημα αυτό και να έχουμε απλώς κάποιους συγκεκριμένου κανόνες για τα συστήματα εξυγίανσης. Χρειαζόμαστε ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες δεν θα έχουν εσωτερικά συστήματα τα οποία τελικά θα παρεμπονδίζουν τα σχέδια εξυγίανσης. γιατί νομίζω ότι αν αρχίσουμε να επιτρέπουμε στις αρχές εξυγίανσης να δίνουν επενδυτικές συμβουλές στις τράπεζες, ενδεχομένω να οδηγηθούμε σε προβλήματα. Στο κείμενό μου προβλέπω διάφορες εναλλακτικέ λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εγκριθούν. Προσπάθησα όμως να είμαι συγκεκριμένο και να τις περιορίσω όσον αφορά τώρα το ζήτημα της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνομαι στον Άλλη Σμιτ και σε άλλους συναδέλφους. Και η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική. Και προσπαθώ να προωθήσω την ιδέα αυτή μέσω αυτής της έκθεσης. Δηλαδή, να φέρουμε την ευθύνη σε ένα κατώτερο επίπεδο, σε επίπεδο των τραπεζών και των μετόχων, να έχουμε ένα πιο αποκεντρωμένο χαρακτήρα, αν θέλετε, στον τομέα της ευθύνης. Και ο αποκεντρωμένος αυτός χαρακτήρας επίσης θα πρέπει να πάει και στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Διαφορετικά οδηγούμε ένα νέο ηθικό κίνδυνο. Θα πρέπει να υπάρχουν πολλές συναλλακτικέ για τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό βλέπουμε και στα πλαίσια του ESF. Εκεί υπάρχει μια πολύ έντονη παρέμβαση του κράτους, η οποία όμως δεν ελέγχεται ουσιαστικά, για την οποία δεν προβλέπονται συγκεκριμένοι νομοθετικοί κανόνε. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι τράπεζε και ότι τα κράτη-μέλη θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη που του αντιστοιχεί και θα πρέπει να δούμε μαζί πώ μπορούμε να καταλήξουμε σε συστήματα αλληλέγγυα. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα εθελοντικό χαρακτήρα και ακριβώ αυτό παρουσιάζω αυτή την έκθεση. Σα ευχαριστώ πολύ. Και κάτι τελευταίο, αν με επιτρέπετε. Πραγματικά προσβλέπω στη συζήτηση που θα έχουμε με τους σκιώδεις ηγητές και με όλους τους άλλους συναδέλφους. Πολλά από τα πράγματα που συζητάμε έχουν μια έντονη τεχνική φύση και σαφώς εγώ διατηρώ ένα ανοιχτό πνεύμα. Πολλά ζητήματα είναι πάρα πολύ τεχνικά, κάποια είναι ιδεολογικά. Πιστεύω πάντως ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό παρανομαστή, ο οποίος θα μας βοηθήσει όλους. Ευχαριστώ Γκούνερ και σε ευχαριστώ για το γεγονός ότι αντιμετωπίζεις και τις συνδέσεις με το, την οδηγία CRD4 και το πώς θα πρέπει να συναρμοστούν αυτά τα δύο νομοθετήματα. Δεν είναι πολύ εύκολο. 28 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίε το μεσημέρι. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε στις 17-18 Δεκεμβρίου να επανέλθουμε στη συζήτηση αυτού του θέματος και των τροπολογιών. Και ο στόχος μας είναι να ψηφίσουμε τον επόμενο Μάρτιο και να έρθουμε στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Θα έχουμε λοιπόν αρκετό καιρό για να κάνουμε τα απαραίτητα και να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Προχωράμε τώρα στο σημείο 9 που είναι τα RIBS, τα έγγραφα πληροφορίας για τα επενδυτικά προϊόντα. Η Υπερβάνς Μπερές είναι η αρμόδια για τα θέματα αυτά και θα τις δώσω στο λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λοιπόν κάνει την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Το κείμενο αυτό βρίσκεται επιτάπητος από τον προηγούμενο τον Ιούλιο. Όλοι οι συνάδελφοι λοιπόν οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στα θέματα αυτά είχαν την ευκαιρία να αναδιευθύσουν το κείμενο αυτό και ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση από λομπίστες, από ομάδες πίεσης, από το εξωτερικό που προσπαθούν να διαμορφώσουν την άποψη σε σχέση με το κείμενο αυτό. Πρόκειται για ένα, μια πρόταση κανονισμού και ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα εργαλείο το οποίο στην αρχή φάνηκε ότι ήταν ιδιαίτερα θετικό, αλλά στη συνέχεια διεφάνει ότι πολλές από τις ρυθμίσεις αυτού του κανονισμού αφορούν ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν από τα κράτη-μέλη, ιδίως σε ό,τι αφορά το καθεστώς των κυρώσεων. Ο στόχος του κειμένου είναι να εξασφαλίσει την προστασία των μικροεπενδυτών με την ε, βασική ιδέα ότι ήδη πριν από την τρέχουσα κρίση αλλά ιδίως και μετά από την έκρηξη της κρίσης είναι απαραίτητο να προστατευτούν οι μικροεπενδυτές γιατί είναι σημαντική η εμπιστοσύνη τους προς τις επενδύσεις για να μπορούν να κινητοποιηθούν οι επενδύσεις τους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Πέραν της ανάγκης προστασίας των μικροεπενδυτών υπάρχουν δύο άλλοι στόχοι οι οποίοι συμπληρώνουν την πρόταση αυτή κανονισμού. Ένας δεύτερος στόχος είναι η εξασφάλιση ίσων συνθήκων ανταγωνισμού. Να υπάρξει λοιπόν μια αντιμετώπιση όλων των προϊόντων που μπορούν να προσελκύσουν τις επενδύσεις των μικροεπενδυτών, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα και χωρίς τρευλώσεις μεταξύ αυτών. Και ένας τρίτος στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι συνθήκες εμπορίας των προϊόντων που απευθύνονται σε μικροεπενδυτές λειτουργούν σωστά. Γι' αυτό το PRIPS φαίνεται ότι είναι ένα πολυκείμενο, ένα κείμενο το οποίο εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους και παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Εγώ έχω δημιουργήσει ένα πίνακα με τη βοήθεια της γραμματείας που δείχνει ποια είναι η κατάσταση σε γραφικό επίπεδο το κείμενο αυτό βρίσκεται στο σταυροδρόμι πολλών άλλων, αν θέλετε, νομοθετικών κειμένων. Συνδέεται με την MIFID, την οδηγία για τα επενδυτικά μέσα, αλλά συνδέεται επίσης και με το κείμενο που αφορά τη διαμεσολάβηση στα, στον, στον χώρο των ασφαλιών. Το πρώτο ερώτημα που πιστεύω ότι θα πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας σε σχέση με την προστασία των επενδυτών είναι η σφαίρα εφαρμογής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε μια σφαίρα εφαρμογής που είναι σχετικά περιορισμένη. Γιατί αναφέρεται στην υποχρέωση των παραγωγών επενδυτικών προϊόντων που αναφέρονται, που απευθύνονται καλύτερα στους μικροεπενδυτές. Είναι υποχρέωση λοιπόν, θέλει να θεσπίσει την υποχρέωση, να δίδουν ένα κέριο έγγραφο πληροφόρησής τους. Είναι όπως πηγαίνει κανείς να αγοράσει ένα πλυντήριο και πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει απλώς ένα διαφημιστικό φυλάδιο, αλλά ένα έγγραφο το οποίο εξηγεί πώ λειτουργεί το πλυντήριο. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να υπάρχει ένα φυλάδιο που δίνει στου επενδυτέ τι απαραίτητε πληροφορίε σε λεπτομεριακό επίπεδο. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι ποια είναι τα επενδυτικά προϊόντα τα οποία πρέπει να καλύπτονται από μια τέτοια ρύθμιση. Εγώ ειλικρινά θα προτιμούσα να καλυφθεί το σύνολο των προϊόντων μικροεπένδυσης και όχι ένα πακέτο. Θα προτιμούσαμε να έχουμε ένα ρίψ και όχι ένα πρίψ, λέει η ομιλήτρια. Αλλά ακόμα και αν περιοριστούμε στα πλαίσια του πρίψ, η οδηγός γραμμή της Κομισιόν ήταν ότι δεν καλύπτονται τα προϊόντα των οποίων η απόδοση συνδέεται μονάχα στο επίπεδο των επιτοκίων ή αυτών που καλύπτονται από άλλα εργαλεία όπως είναι τα προσπέκτους, τα διαφωτιστικά φυλάδια. Αν σκεφτούμε τώρα τι θέλει να κάνει η Κομισιόν και συμφωνούμε με αυτό, ε, προστασία των μικροεπενδυτών, ε, συνθήκες εμπορίας των προϊόντων αυτών, ισότης ανταγωνισμού, Πιστεύω ότι θα πρέπει να κανει η κομισιον και συμφωνουμε με αυτο προστασια των μικροεπενδυτων ε συνθηκες εμποριας των προιοντων αυτων ισοτητας ανταγωνισμου πιστευω οτι θα πρεπει να ζητησουμε μια διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής αυτού του νομοθετήματος για τρία κυρίως είδη προϊόντα που είναι οι μετοχές και τα εργαλεία δημοσίου χρέους, ομολόγια, ομολογίες δημοσίου χρέους, γιατί δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι όλα τα προϊόντα που καλύπτουν από ένα προσπέκτους έχουν χαρακτήρα ισοδύναμο. Για ένα μικρό επενδυτή υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες ε, αναγνωσιμότητας αυτών των φυλαδίων ένα δεύτερο είδος προϊόντων για τα οποία πρέπει να διευρύνουμε τη σφαίρα εφαρμογής είναι ορισμένα τραπεζικά προϊόντα. με διαφορετικά είδη ε, τόκων που δίνουν ή άλλων προϊόντων. Και επίσης είναι τα τα προϊόντα <clears throat> ασφάλειας ζωής τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ανεξάρτητα λοιπόν από το γεγονός ότι η Κομισιό θέλει να καλύψει συνολικά όλα τα προϊόντα της λεγόμενης λιανικής αγοράς επενδύσεων, αν έχουμε αυτό το κέριο έγγραφο, το έγγραφο κλειδί για τις επενδύσεις όπως αναφέρεται, μονάχα για τα προϊόντα για τα οποία θέλει η Κομισιόν να υπάρξει αυτή η κάλυψη, κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου ο μικρός επενδυτής, ο οποίος δεν γνωρίζει πολλά για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, θα χρησιμοποιεί για την ενημέρωσή του το πιο ευανάγνωστο έγγραφο, <clears throat> το οποίο θα καλύπτει τα πιο πολύπλοκα προϊόντα στα οποία έχει πρόσβαση. Θα πηγαίνει λοιπόν στις ε, καταθέσεις ε, που στα από τα ταμιευτήρια θα πηγαίνει σε αυτά τα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από την πρόταση της Κομισιόν. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να σας αναφέρω. Είναι και το περιεχόμενο αυτό του εγγράφου κλειδί. Πού αναφέρονται, παραδείγματος χάρη, οι ενδείξεις κινδύνου και με ποιο τρόπο ε, παρουσιάζεται ο κίνδυνος αυτών των επενδύσεων. Αυτό το οποίο περιέχεται αυτή τη στιγμή ως ένδειξη κινδύνου είναι ένας δείκτης ο οποίος κοιτάζει προς τα πίσω ουσιαστικά. Είναι σαν να είναι ο κίνδυνος ο ο κίνδυνος να προέρχεται από το παρελθόν, ενώ ο κίνδυνος προέρχεται από το μέλλον. Αν βλέπουμε μονάχα την απόδοση στο παρελθόν όλων αυτών των ε, μέσων επένδυσης, κινδυνεύουμε να υποτιμήσουμε το μελλοντικό κίνδυνο. Ε, τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από την εξέλιξη της ρευστότητος ή από τους κινδύνους αντισυμβαλωμένων κτλ. Επομένως θα πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη συζήτηση για να δούμε τι μορφή θέλουμε να έχουμε για τους δείκτες κινδύνου. Ένα τρίτο σημείο ανησυχία αφορά τη φύση των επενδύσεων. Πιστεύω προσωπικά ότι χωρίς τώρα να θέλουμε να δίνουμε ένα κοινωνικό χαρακτήρα ή ένα περιβαλλοντικό χαρακτήρα στα πάντα, μας ενδιαφέρει να ξέρουμε και πού θα επενδυθούν τα χρήματα αυτά τα οποία προέρχονται από τους μικροεπενδυτές. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και για λόγους διδακτικούς και για να αντιμετωπίσουμε τις όλο πιο έντονες ανησυχίες των επενδυτών θα είναι χρήσιμο να αναφέρεται αυτό στο έγγραφο κλειδί. Ένα τέταρτο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η γέφυρα μεταξύ του εγγράφου κλειδί και του εγγράφου που αφορά τη, τα μέσα επενδύσεων σε κινητές αξίες. σεκα. Ξέρουμε ότι τα έγγραφα αυτά, τα πληροφοριακά, καλύπτουν περισσότερα προϊόντα από τα ΟΣΕΚΑ και μόνο. Η Κομισιόν έχει προβλέψει λοιπόν αυτή την γεφύρωση προς τα έγγραφα αυτά. Πώς ακριβώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, πώς θα συμπεριλάβουμε τα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από ευρύτερα έγγραφα ακόμα και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική πρόταση. Πέμπτη ανησυχία. Το θέμα των κυρώσεων. και του καθεστώτος το οποίο πρέπει να διέπει τα προϊόντα τα οποία έχουν για τα οποία έχει διακριβωθεί ότι περιλαμβάνουν κινδύνους. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία δυσκολία και η οποία μας υπενθυμίζει αυτά τα οποία ψηφίσαμε στο παρελθόν στο νομοθέτημα ΜΙΦ, όπου αναφερόμαστε κυρίως στις εξουσίες της ε, αρχής για τις ε, αγορές αξιογράφων. Ενώ εδώ θα έχουμε μια άλλη εποπτική αρχή που θα είναι, δεν θα είναι η αρχή για τα αξιόγραφα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ένα ισότιμο επίπεδο προστασίας. Δύο ακόμα σημεία για τα οποία θα ήθελα να αναφερθώ και θα περιμένα και εδώ τις προτάσεις των συναδέλφων. Καταρχήν, το έγγραφο αυτό το οποίο προέρχεται από τον παραγωγό ενός επενδυτικού εργαλείου και στη συνέχεια δίνεται από αυτόν ο οποίος διανέμει αυτά τα προϊόντα επενδύσεων. Ο στόχος του κειμένου όμως αυτού είναι ουσιαστικά να πληροφορήσει τον μικροεπενδυτή. Εγώ δεν έχω τώρα αριθμητικά στοιχεία να σας παραθέσω, αλλά διαισθητικά και μετά από συζητήσεις που έχω κάνει με πολλούς συναδέλφους, Ξέρω ότι για ένα μικροεπενδυτή αυτό το οποίο έχει σημασία για μια επένδυση είναι οι συμβουλές που θα πάρει από κάποιον. Είναι κάτι το οποίο είναι αποφασιστικό. Οι συμβουλές που παίρνει είναι αυτές οι οποίες προσδιορίζουν κατά το 1 τρίτο τουλάχιστον τις ε, επιλογές του. Ένα δεύτερο τρίτο έχει να κάνει με το φορολογικό καθεστώς το οποίο υπόκειται το προϊόν αυτό λιανικών επενδύσεων. Είναι αποφασιστικού χαρακτήρα και το φορολογικό καθεστώς. Και βλέπω τώρα εγώ όλα αυτά τα διαφημιστικά, τα οποία έχουν πολύ ωραία χρώματα κτλ. που λένε ενδιαφέροντα πράγματα για τον επενδυτή. Αλλά αν δεν υπάρχει και κάποιο κείμενο το οποίο να εξηγεί ποιο είναι το φορολογικό καθεστώς το οποίο ε, αφορά αυτό το επενδυτικό προϊόν είναι ελλειπής η πληροφόρηση. Δεν ανταποκρίνεται κανείς στις ανησυχίες των μικροεπενδυτών. Θα ήθελα λοιπόν να προβλέπετε ότι υπάρχει κάποιο κομμάτι της σελίδας όπου θα πρέπει αυτός ο οποίος διανέμει το προϊόν αυτό να συμπληρώσει το φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τα προϊόντα αυτά. Και ένα τελευταίο θέμα είναι φυσικά το καθεστώς το οποίο υπόκειται τα προϊόντα από τρίτες χώρες και θα πρέπει εδώ να εξετάσουμε κατά πόσον αυτός ο, ο κατάλογος υποχρεώσεων περιλαμβάνει και προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες. Αυτά. Um, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, εκ μέρους του ΕΛΚ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι ο αρχικός στόχος αυτής της ε, νομοθεσίας ε, για τα ΠΡΙΠ ε, είναι δικαιολογημένος. Χρειαζόμαστε καλύτερη προστασία, καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και χρειαζόμαστε επίσης σαφέστερους και περιεκτικότερους κανόνες για να μπορούμε να συγκρίνουμε τα διάφορα προϊόντα. Κατά τα άλλα, όσον αφορά σε αυτή την πρόταση της Επιτροπής, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που έθιξε η συγκήτρια, με τα οποία συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι έχουμε βέβαια ακόμα ε, αρκετή δουλειά μπροστά μας για άλλου είδους θέματα. Να πω το εξής πρώτα απ' όλα. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε τη συγκρισιμότητα και την ικανοποιητική ενημέρωση του καταναλωτή και την εύκολη πρόσβασή του σε ενημέρωση, αυτό εύκολα λέγεται, δύσκολα γίνεται. Και ένα από τα πράγματα που με ανησυχούν είναι ότι υπάρχει αρκετά ε, πρόσφατη νομοθεσία για τους οσεκα Είναι μόλις τώρα τελευταία που ε, θεσπίστηκε η, η νομοθεσία αυτή. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω η ΟΣΕΚΑ και τα ΠΡΙΠ να αναφέρουν στην ίδια γραμμή. Γιατί αλλιώς ελοχεύει ο κίνδυνος οι καταναλωτές τουλάχιστον στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα αλλά και ε, μακροπρόθεσμα να κατακλείζονται από δύο ε, διαφορετικές δέσμες ε, πληροφοριών. Και δεν είμαι σίγουρη, καθόλου, μα καθόλου σίγουρη κατά πόσον αυτό θα εξυπηρετήσει τον τελικό σκοπό. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα χρησιμοποιούνται καλύτερα οι ΟΣΕΚΑ στη δική μας την περίπτωση. Τώρα πάμε στα ε, προϊόντα ασφαλιστικών επενδύσεων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα, ασφαλιστικά προϊόντα, ε, τα οποία ε, είναι στην ίδια κατεύθυνση όπως και τα άλλα προϊόντα, λιανικά προϊόντα επενδύσεων. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε τη συγκρισιμότητα. Εγώ δεν έχω την απάντηση δυστυχώς, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε διεξοδικότερα το θέμα αυτό. Και πάμε τώρα στο εύρος. Ξέρω ότι τα συνταξιδοτικά ταμεία δεν περιλαμβάνονται κυρίως στις κανονικές συντάξεις. Ε, όμως ε, νομίζω ότι ε, πρέπει να αποφασίσουμε Μήπως θα πρέπει και αυτά, αυτές οι ε, κατοχυρωμένες συντάξεις ε, θα πρέπει να επενδύονται ή όχι. Τώρα, ένα πρόβλημα που έχω είναι το εξής. Ε, ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται ο κίνδυνος. Εγώ προσωπικά έχω κάποιες επιφυλάξεις ε, για το κατά πόσον θα έπρεπε αυτό το έγγραφο για τα ΠΡΙΠ να είναι αυτοτελές, να είναι μόνο του και να προσφέρει αυτό τις ε, πληροφορίες ε, στον καταναλωτή. Βασικά στην αξιοδοτικά Ναι. Το θέμα είναι ε, κατά πόσον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το απλό σύστημα επιμερισμού των κινδύνων ε, ίσως ε, όμως με τον τρόπο αυτό να παραπλανήσουμε τους επενδυτές Αυτοί δηλαδή μπορούν να πιστέψουν ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι πιο σταθερό και τουλάχιστον επιδεικνύει ένα ιστορικό κερδοφορίας, τότε και ο επενδυτής ε, να σκεφτεί ότι αυτή είναι ε, λιγότερο επικίνδυνη επένδυση. Ε, το θέμα είναι βέβαια και η δομή του κόστους. Ο επενδυτής ίσως τελικά χάσει τα χρήματά του, όχι λόγω της μεταβλητότητας του προϊόντος, αλλά λόγω της διάθρωσης ε, του κόστους που μπορεί να οδηγήσει στο να μην κερδίσει τίποτα τελικά από την επένδυσή του, ακόμα και αν εξαφανιστεί ο κίνδυνος της ε, μεταβλητότητας. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτούς τους ε, δείκτες γιατί ενδέχεται να παραπλανήσουν τους καταναλωτές ε, ως προς την κατανόηση του προϊόντος. Να καταλάβουν ότι υπάρχει κίνδυνος να μην κερδίσουν από αυτή την επένδυση και σε ορισμένες περιπτώσεις ε, η απόδοση να είναι χαμηλότερη του πληθωρισμού. Μόνο δηλαδή εκείνος που πουλάει κερδίζει. Αυτό Αυτά είναι τα βασικά θέματα και ίσως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, διαφορετικά σενάρια και διαφορετικά στοιχεία. Κατόπιν, υπάρχουν ορισμένα θέματα στην εποπτεία, α, εποπτεία αν θα επεκταθεί αυτή και στις ε, συντάξεις. Ε πρέπει να υπάρχει μια επαφή με τον καταναλωτή, κυρίω όσον αφορά την προστασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται εγώ είμαι η εκπρόσωπος της Άλντε. Θα κάνω τα σχόλιά μου από εδώ. Όσον αφορά το ζήτημα το οποίο έθιξες, ε, Περβάνς, και εγώ συμφωνώ μαζί σου, ιδίως όταν εξετάζουμε συνταξιοδοτικά προϊόντα, για τα οποία τα κράτη-μέλη λένε «Κοιτάξτε, δική μας στάση είναι διαφορετική από ό,τι είναι σε κάποια άλλα κράτη». Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει έστω μία κάποια συγκρισιμότητα στα προϊόντα αυτά και να έχουμε και κάποια πιο απλά προϊόντα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βλέποντας εδώ πέρα τις δύο εξαιρέσεις, δηλαδή όταν η απόδοση έχει να κάνει μόνο με τα επιτόκια και αυτό όμως καταλαβαίνεις ότι μπορεί να καλύπτει κάτι το ιδιαίτερα πολύπλοκο. Νομίζω λοιπόν ότι ο μικροεπενδυτής ενδεχομένως να χρειάζεται έστω και μια κάποια απλή καθοδήγηση και στην περίπτωση αυτή. Όταν τώρα η πληροφόρηση αυτή καλύπτεται από κάποιο άλλο βασικό κείμενο πληροφόρησης, τότε θα πρέπει να καταφέρνουμε κάπως να συνδυάζουμε αυτά τα δύο κείμενα, προκειμένου να αποφύγουμε αντιφάσεις. ή να αποφύγουμε σωστικά να παραπλανήσουμε ή να αποσυντονίσουμε τον μικροεπενδυτή που, στον οποίο θα λέμε να κοιτάει πολλά διαφορετικά κείμενα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και μία εξήγηση όσον αφορά το φορολογικό καθεστώς του προϊόντος, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για τους ε, επενδυτές, οι οποίοι ε, προσπαθούν να αποτιμήσουν το ρίσκο το οποίο διατρέχουν στα πλαίσια της αγοράς. Και το ρίσκο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ο κίνδυνος αυτός διαφοροποιείται με βάση το φορολογικό καθεστώς το οποίο προβλέπεται για το επενδυτικό προϊόν. Πρέπει λοιπόν και αυτό κάπως να το εξηγήσουμε. Αναφέρθηκες επίσης στην αγορά ενός ψυγείου. Μα ξέρεις ότι όταν αγοράζεις ένα ψυγείο, τουλάχιστον τα πήγα εγώ να αγοράσω ένα ψυγείο, είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά για παράδειγμα την κατανάλωση ενέργειας και το καθεξής. Άρα νομίζω ότι ε, είναι πολύ δύσκολο το να καταφέρνουμε να παρέχουμε ισότιμα όλες τις πληροφορίες. Ενδεχομένως να πρέπει να γίνει μια κάποια διάκριση στις πληροφορίες αυτές και καταλαβαίνετε πόσο πιο πολύπλοκα γίνεται τα πράγματα όταν πρέπει να δοθούν πληροφορίες για ένα επενδυτικό προϊόν. Όσον αφορά το ζήτημα της ε, απλοποίησης. Ζήτημα το οποίο με έχει απασχολήσει πάρα πολλέ φορέ στο παρελθόν. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Α μην υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα σε σημείο που δεν σημαίνουν πλέον τίποτα, δεν δίνουν καμία πληροφόρηση. Αλλά α αποφύγουμε και την άλλη κατάσταση, την άλλη πλευρά, όπου θα δίνουμε πάρα πολύ λεπτομερεί και τελικά παραπλανητικέ πληροφορίε. είναι πάρα πολύ σημαντικό το επενδυτικό προϊόν να συνοδεύεται από ισορροπημένες πληροφορίες που θα δίνουν την απαραίτητη ενημέρωση στο μικροεπενδυτή. Θα πρέπει οι μικροεπενδυτές χρησιμοποιώντας πληροφορίες αυτές να μπορούν να κάνουν τη σωστή απόφαση, να επιλέξουν το σωστό προϊόν. Πολλές φορές όμως, αν η πληροφόρηση είναι πάρα πολύ εκτενή, αν προβλέπονται πάρα πολλές εξαιρέσεις, αυτό μπορεί με τη σειρά του να αποσυντονίσει τελικά τον μικροεπενδυτή. Μπορεί ο μικροεπενδυτής να μην είναι σε θέση να καταλάβει τελικά που έγκυται ο κίνδυνος. Όσον αφορά τώρα την ενημέρωση των KID, των βασικών εγγράφων πληροφόρησης. Η ενημέρωση αυτή, η αναθεώρηση είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Εγώ Προσωπικά έχω επενδύσει σε διάφορα παιδευτικά προϊόντα και νομίζω ότι ε, πολλές φορές κουράζομαι από το γεγονός ότι μου έρχονται όλο και περισσότερες πληροφορίες. Ε, ξέρετε ότι ε, καταφθάνει ο ταχυδρόμος πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα φέροντας γράμματα τα οποία περιέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Και δεν ξέρω τελικά πιο ποσοστό της σύνταξής μου κατηναλώνεται μόνο και μόνο στην δημιουργία όλων αυτών των έγγραφων πληροφοριών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε σαφώς ενημέρωση της πληροφορίας, επικαιροποίηση της πληροφορίας, όταν όμως αυτό κρίνεται αναγκαίο και να αποστέλνουμε τελικά την ενημέρωση αυτή, να την καθιστούμε διαθέσιμη όταν τη χρειάζεται πραγματικά ο μικροπενδυτής. Και ουσιαστικά να γίνεται αυτή η επικαιροποίηση όταν έχουμε σημαντικέ ουσιώδει αλλαγέ. Πρέπει να δούμε πώ θα καταφέρουμε να το καθορίσουμε το κριτήριο αυτό στα πλαίσια του κειμένου. Εγώ δεν θα ήθελα πάντω να λαμβάνω συνεχώ ενημερώσεις οι οποίες τελικά είναι δαπανηρές και τελικά κατακλείζομαι από πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες δεν καταφέρνω ποτέ να διαβάσω. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να έχουμε κάποια βασικά έγγραφα ενημέρωση, τα οποία όμω να λειτουργούν και στην πράξη. Όσον αφορά τώρα τον κίνδυνο Σαφώς θα πρέπει να προβλέψουμε επιμέρους κεφάλαια που να εξηγούν τους κινδύνους τους οποίους είναι εκτεθειμένος ένας μικροεπενδυτής. Αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα αποφάσεις μας θα πρέπει να συνάδουν με τα όσα προβλέπονται στα πλαίσια των ΟΣΕΚΑ. Όσον αφορά τώρα τα τέλη, το κόστος. Είναι καλό να γνωρίζει ο μικροεπενδυτής ότι το προϊόν το οποίο έχει αγοράσει είναι εκτεθειμένο σε κινδύνους της αγοράς και θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ο επενδυτής ότι πολλές φορές μπορεί το προϊόν το οποίο έχει επιλέξει στην αγορά να αποκτήσει μεγάλη αξία, αλλά αυτή η υπεραξία τελικά δεν θα καταλήξει ποτέ στα χέρια του μικροεπενδυτή και τελικά θα αναλωθεί σε ε, δαπάνες, σε τέλη τα οποία πρέπει να, κατα... καταβάλει ο μικροεπενδυτής. Ο μικροεπενδυτής πρέπει να γνωρίζει τελικά τι καταλήγει στην τσέπη του. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σαφείς παρουσιάζοντας όλη αυτή την αλυσίδα από την λειτουργία και τις επιδόσεις ενός προϊόντος στην αγορά μέχρι τη στιγμή που το προϊόν αυτό φτάνει στα χέρια του μικροεπενδυτή. Πρέπει να γνωρίζει λοιπόν ο μικροεπενδυτής ακριβώς τι θα κερδίσει στο τέλος. Πολλές φορές θεωρεί ότι επιλέγει ένα επικίνδυνο προϊόν το οποίο όμως θα το αποφέρει πολύ μεγάλες επιδόσεις στην αγορά και τελικά απογοητεύεται όταν βλέπει ότι τα χρήματα τα οποία φτάνουν στα χέρια του είναι λιγοστά θα σκεφτώ όλα αυτά τα ζητήματα, θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Αυτή τη στιγμή εξέφρασα κάποιες πρώτες σκέψεις. Ο Σβέν δεν είναι εδώ, γιατί όπως είπαμε είναι πατέρας ή σύντομα θα γίνει πατέρας. Δεν έχω ενημερωθεί ακόμα για το πού βρίσκονται τα πράγματα. Φιλίππα, θα τον εκπροσωπήσεις εσύ. Und ich werde nicht auf Deutsch δεν είμαι ο Σβέν Γίγκολτ, ούτε καν θα μιλήσω στα γερμανικά. Και δεν μπορώ να αναφερθώ στο θέμα του, της γένας, απλώς μπορώ να παίξω το ρόλο της ΜΕΑ σε ό,τι αφορά τη συζήτηση. Μα δεν σκεφτήκατε Σάρων, για το θέμα αυτό. Όλα αυτά που είπες τα λες ότι τα είπες χωρίς να σκεφτείς και τώρα θα σκεφτείς περισσότερο. Σίγουρα ξέρεις τα πράγματα πολύ καλύτερα από ότι εγώ ίδιος αλλά εγώ συμμερίζομαι πολλά από αυτά που είπες. Συγγνώμη που καθυστέρησα όμως να το στην αρχή της ομιλίας σου. Σίγουρα συμφωνούμε και εμείς με την πρόταση της Κομισιόν ότι είναι απαραίτητε οι προσπάθειες για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια προς τους καταναλωτές και τους μικροεπενδυτές που είναι και ο κύριος στόχος αυτού του νομοθετήματος. Υποστηρίζουμε επίσης και το θέμα των κυρώσεων γιατί τον υπάρχουν κανόνες χωρίς κυρώσεις. Αυτό είναι τίγρης με πύληνα πόδια ή χάρτινες τίγρης, σε μας περιπτώσει, και γι' αυτό είναι πολύ θετικό ότι η Κομισιόν υποστηρίζει αυτές τις ε, κυρώσεις. Πού μπορούμε να βελτιώσουμε τώρα αυτό το κείμενο. Ξέρετε ότι εμείς υποστηρίζουμε να υπάρξει μια μετάβαση της οικονομίας προς την κατεύθυνση της πράσινης οικονομίας και εδώ δεν θέλουμε να υπάρξει μια κατά κάποιο τρόπο ε, παραπλάνηση του κοινού με το πρόσχημα της πράσινης οικονομίας. Θέλουμε να υπάρχουν σαφή κριτήρια τα οποία περιέχονται σε αυτό το έγγραφο κλειδί σε σχέση με τον περιφαλλοντικό ή κοινωνικό χαρακτήρα των επενδύσεων. Επίσης, θα θέλαμε να υπάρχει μια καλύτερη εξέταση της καταλληλότητας των προϊόντων που απευθύνονται σε μικροεπενδυτές. Να υπάρχει μια εκ των προτέρων εξέταση της καταλληλότητας αυτών των προϊόντων επομένως να υπάρξει μια προηγουμένη εξέταση αυτών των προϊόντων που να είναι στεναρή, εξάντε πάντα. Επίσης, το γεγονός ότι, ότι ο επενδυτής θα πρέπει να αναφέρει επισήμως ότι έχει διαβάσει και καταλάβει το έγγραφο, θα πρέπει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, ακόμα και αν γίνεται αυτή η επικοινωνία μέσω του ίντερνετ εξ αποστάσεως. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε βέβαια ότι ο επενδυτής θα διαβάσει το κείμενο, θα μπορούσε να το διαβάσει στο διαδίκτυο, αλλά να υπάρχει αυτή η απέτηση. Θα θέλαμε επίσης να υπάρχουν και προβλέψεις για μελλοντικέ εξελίξεις του προϊόντος. Από ό,τι βλέπω η πρόταση Κομισιόν καλύπτει τις συντάξεις για τα θέματα αυτά, τα συνταξιοδοτικά προϊόντα Ίσως αυτός ο δείκτης όμως θα πρέπει να αφορά και άλλα μακροχρόνια προϊόντα επενδύσεων, να αναφέρει το γενικό, το κεντρικό σενάριο και να αναφέρει και την ευαισθησία αυτού του σενάριου σε διάφορες εξελίξεις και τι θα μπορούσε να προκύψει. Για τα προϊόντα που έχουν απεριόριστη διάρκεια για τα προϊόντα αυτά τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει και κάποια εκτίμηση για την διάρκεια του προϊόντος αυτού, αν δεν είναι καθορισμένο εκ των προτέρων. Και επίσης για την εκτίμηση του κινδύνου. Θα θέλαμε να υπάρχει και κάποιος δείκτης ο οποίος να περιλαμβάνει όχι μόνο τον κίνδυνο αγοράς αλλά και τον κίνδυνο αντισυμβαλωμένων και τον κίνδυνο ρευστότητος που πολλές φορές είναι πιο σημαντική από τον κίνδυνο ε, αγοράς. Διαδικασίες θεραπείας, εξοδικαστικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών και αυτό θα πρέπει να το δούμε στο έγγραφο. Υπάρχουν ορισμένε περιοχές για τις οποίες θα πρέπει να υπάρξει μια διεύνηση της πρότασης, όπως παραδείγματος χάρη, να καλύψει η πρόταση αυτή και τον σχεδιασμό των προϊόντων γιατί η τωρινή νομοθεσία για τα προϊόντα αυτά δεν είναι πλήρης. Επίσης να παρουσιάσετε το συνολικό κόστος προς τον καταναλωτή σε επίπεδο νομισματικό και συγκεκριμένο, να καταλαβαίνει δηλαδή ο καταναλωτής τι θα πληρώσει συνολικά, ενδεχομένως και μία ε, εκτίμηση <clears throat> της ε, απόδοσης αυτού του προϊόντος και μία σύγκριση με ένα συγκρίσιμο ασφαλές προϊόν αντίστοιχης ε, Διάρκεια ορίμανσης, παραδείγματος χάρη κρατικά ομόλογα. Και επίσης <clears throat> όταν παρουσιάζεται η απόδοση επί τη βάση ιστορικών σενάριων θα πρέπει να δείχνεται με γραφικά αυτή η εξέλιξη ώστε να είναι κατανάλωση. Αυτά είναι τα βασικά λοιπόν στοιχεία που ήθελα να σας μεταφέρει ο συνάδελφός μου ο Σβέν εάν δεν κολλιόταν και ελπίζω ότι το έκανα με έναν τρόπο που θα σας Thank σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ε, φαντάζομαι όλα ε, θα χαίρεται πάρα πολύ που θα ε, υπάρξει αυτό το νέο παιδί, kid, γίνεται ένα λογοπαίγνιο εδώ. Ζητώ συγγνώμη από όλου βέβαια που δεν καταλαβαίνουν ε, αυτό το δικό μου το λεπτό χιούμορ που είναι βέβαια και δύσκολο να μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα από τα αγγλικά. Εν πάση περιπτώσει, ε, θεωρώ ότι είναι ε, σημαντικό το ότι έχουμε κάνει εμπειρία με τους ΣΕΚΑ. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής. Θα πρέπει να είμαστε σαφέστεροι αυτό το KID. Τελικά τι θα κάνει, θα υπάρχουν ασφαλέστερα προϊόντα, θα είναι πηγή πληροφοριών ή θα είναι και τα δύο. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι από αυτού ποιες είναι οι προθέσεις μας, ε, αν θα είναι ένα προσυμβασιακό ε, αντικείμενο. Επίσης, ε, θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει παραπλάνηση. Αλλά θα πρέπει και οι πληροφορίε που δίνονται να είναι σαφεί. Και ένα τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να επιτρέπουμε στους επενδυτές να αποκτούν περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά το θέμα της αστικής ευθύνης, ε, νομίζω εκεί πρέπει να υπάρχουν ε, περισσότερες λεπτομέρειες, ε, όπως και σε σχέση με τους ΣΕΚΑ. Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι κατά πόσο οι ανησυχίες που υπάρχουν είναι νομιμοποιημένες ή όχι. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι το έγγραφο αυτό, το KID, δεν πρέπει θα να αντιμετωπίζεται ως το μόνο έγγραφο που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο επενδυτής ε, για την επένδυσή του. Και θα πρέπει βεβαίω να υπόκειται και σε καθεστώς ε, αστικής ευθύνη. Αν δούμε λοιπόν τις αναταραχές ε, στα συνταξιδοτικά συστήματα των κρατών μελών, στη δική μου τη χώρα, παραδείγματος χάρη, μερικοί τώρα δεν επιλέγουν να μπουν σε ένα ασφαλιστικό ταμείο, απλά τους πιέζουν να μπουν με το ζόρι. Γι' αυτό λοιπόν ε, καταλαβαίνετε ότι πρέπει και ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συζητηθεί το θέμα των συντάξεων ε, και προτιμώ να γίνει αυτή η κουβέντα πριν προχωρήσουμε πιο κάτω. Τώρα, όσον αφορά τις ε, εναλλακτικέ λύσεις ε, διαμεσολάβησης, ε, κατά πόσον μπορεί να είναι ταχύτερη η αποζημίωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές διατάξεις από, την από αυτές που ήδη ισχύουν στην κείμενη οδηγία. Όσον αφορά τώρα το να ανοιχτεί το πλαίσιο για να συμπεριληφθούν όλα τα επενδυτικά προϊόντα, το κατανοώ αυτό, όμως πρέπει να δούμε μήπως απομακρυνόμεθα από την αρχή, αρχικό κείμενο αυτό το KID. Και έχοντας ακούσει αυτά που είπε η κυρία Μπερές, πρέπει να σας πω, κατανοώ αυτά που λέει, αλλά μίλησε πραγματικά για κρατικό και ή δημόσιο χρέος. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει ενδιαφέρον ε, αυτό το KID για το ελληνικό δημόσιο χρέος. Πάντως, ακόμα και σήμερα, οι περισσότεροι καταναλωτές όταν ε, τοποθετούν ε, τα χρήματά τους ε, στην τράπεζα πιστεύουν ότι παραμένουν εκεί και όποτε θέλουν μπορούν να τα πάρουν πίσω. Ενώ η αλήθεια είναι, τα βάζει στην τράπεζα, η τράπεζα τα δίνει περαιτέρω, δίνει πίστη, Γι' αυτό λοιπόν οι καταναλωτές ε, θα πρέπει να γνωρίζουν ε, ποιες είναι οι ε, εξασφαλισμένες καταθέσεις, ποιοι είναι οι δεσμευμένες καταθέσεις, οτιδήποτε. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι κατά πόσον πρέπει όλα αυτά να γίνουν εδώ ή ενδεχομένως σε άλλο χώρο μαζί με την εισηγήτρια και τους σκιώδης εισηγητές. Σε γενικές γραμμές όσον αφορά την προστασία των επενδυτών πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί ο συνήθως ε, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Καλύτερα λοιπόν οι πληροφορίες που δίνουμε είναι να είναι κατανοητές, να μην τους κατακλίζουμε, τους ε, ε, καταναλωτές γιατί υπάρχει και το πρόβλημα ότι ε, πολλές φορές ο καταναλωτής ε, δεν διαβάζει όλες αυτές τις πληροφορίες που τα αποστέλνουν. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκολας δεν είναι παρόν. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο. Η Κέιτ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. ως σκιώδης εισηγήτρια στο MIFID, στο παρελθόν και στο MIFIR, θέλω να τονίσω ότι σίγουρα συνδέεται αυτή η, αυτό το νομοθέτημα με προηγούμενες οδηγίες. Και η συζήτηση για ζητήματα από το πρίψη είχε πολιτικοποιηθεί ιδιαίτερα. Και φοβάμαι ότι η συζήτηση αυτή δεν εστιάζεται στις ανάγκες του καταναλωτή όπως τα περίμενε κανείς. Θα ήθελα λοιπόν αυτό το έγγραφο να εστιάζει στις ανάγκες του καταναλωτή και να παίζει το ρόλο της προστασίας των καταναλωτών και μικροεπενδυτών εναντί των αποφάσεων που θα πάρουν. Δεν νομίζω ότι έχουμε επιτύχει τη σωστή ισορροπία στις προηγούμενες συζητήσεις και τα πράγματα θα είναι ίσως ακόμα πιο μπερδεμένα στους τριγωνικούς διαλόγους και δεν θα προστατεύουν τόσο πολύ τον καταναλωτή. Ένα από τα συμπεράσματα των προηγουμένων συζητήσεων είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια υποχρέωση με ένα τυποποιημένο τρόπο να αναφέρονται όλα τα πρόσθετα κόστη και τέλη που έχει να υπομειστεί ο καταναλωτής και ο μικροεπαιδητής. Πρέπει να το εξασφαλίσουμε λοιπόν και στο έγγραφο KIT, στο έγγραφο για το κομβικό αυτό έγγραφο και επίσης η συγκρισιμότητα μεταξύ των προϊόντων είναι κάτι το πολύ δύσκολο αλλά είναι απαραίτητο. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που για ένα ε, επενδυτικό προϊόν υπήρχαν 12 είδη χωριστών τελών και πρόσθετων ε, καταβολών που γίνονται από τον επενδυτή. Δεν πρέπει λοιπόν κανείς να μπαίνει σε μια τέτοια σύμβαση χωρίς να ξέρει τι ακριβώς θα πληρώσει συνολικά. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και να βοηθήσουμε τον μικροεπενδυτή να καταλάβει τι πρόκειται. Και φυσικά η αγορά δεν θέλει να αποκαλύψει όλα αυτά τα πρόσθετα τέλη, τις πρόσθετες καταβολές. Πρέπει να τους υποχρεώνει το νομοθέτημα αυτό. Και επίσης πρέπει να υπάρξει και μια συνέχεια μεταξύ των προηγουμένων προϊόντων και ε, νομοθετημάτων και του τρέχοντος νομοθετημάτων γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει να υπάρξει μια πλήρης συγκρισιμότητα. Οι μικροεπενδυτές δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά μεταξύ διαφόρων είδων, προϊόντων και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Αν δεν το κάνει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κανείς άλλος δεν θα ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα. Λόγω και του θέματος των επί των προβλημάτων επικουρικότητας για τα επενδυτικά θέματα και το είδαμε αυτό και στις συζητήσεις για τη ΜΥΦΙΤ. Τα κράτη-μέλη <clears throat> μπορούν, μπορούν να εφαρμόσουν τις ε, οδηγίες με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι διακριτικός. Για το θέμα αυτό θα πρέπει όμως για το έγγραφο αυτό το κομικό έγγραφο θα πρέπει να ξέρουν ποιος είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας για την εποπτεία όχι μόνο του χρηματοπιστωτικού αυτού προϊόντος, αλλά και του φορέα που πουλάει αυτό το προϊόν. Για αυτούς τους λοιπόν τους ε, για αυτές τις χώρες και τους δημιουργικούς φορείς που εφαρμόζουν απαγόρευση για ορισμένα προϊόντα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα, στις χώρες αυτές θα ξέρουν αν οι άλλες χώρες ε, εφαρμόσουν τέτοιου είδους απαγορεύσεις και επομένως ποιο είναι το επίπεδο προστασίας του οποίου απολαμβάνουν και εγώ ξέρω από δική μου εμπειρία, γιατί όταν η μητέρα μου αγόρασε ένα προϊόν συνταξιοδοτικού χαρακτήρα, τη ζήτησα να ρωτήσει αν ο σύμβουλος για τις επενδύσεις ήταν υποκείμενος σε κάποια εποπτεία και φαίνεται ότι δεν υπέκειτο στις εποπτικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρει ο μικροεπενδυτή όλα αυτά τα στοιχεία και γι' αυτό το, η πρόταση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για το κέριο έγγραφο και θα πρέπει να του καλύπτει περισσότερο στι ανησυχίε του από ό,τι προηγούμενα έγγραφα. Αν δεν θέλει κανένα άλλο. Νομίζω ότι αυτό που είπε η ΚΕΙ, ξέρουμε ότι όταν κάναμε την οδηγία, αντιμετώπισαν την οδηγία για τις, πληρω... για τις υπηρεσίες πληρωμών, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρεται ποιος είναι ο κάθε επόπτης για τις, ε, σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις. Ήταν σημαντικό να ξέρει ο καταναλωτής ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι αρμόδιος ρυθμιστής όταν γίνεται μια πρόταση προς κάποιον να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό. Πρέπει όλα αυτά λοιπόν να εμφανίζονται με σαφή τρόπο στο φυλάδιο. Θέλει κάποιος άλλος λοιπόν να λάβει το λόγο στο θέμα αυτό. Εντάξει, επανέρχομαι στην Περβάνος τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ξεκινάει καλά η συζήτηση αυτή. Βλέπω ότι υπάρχουν και δυνατότητες σύγκλησης των απόψεών μας σε διάφορα σημεία όσον αφορά τη συγκρισιμότητα. Όλοι έχουμε κατά νου αυτό το στόχο. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε πολύ στενά, συγκεκριμένα και με την IMD, προκειμένου να καταφέρουμε να συντονίσουμε το κείμενο αυτό και με το άλλο το κείμενο, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έχει παρουσιάσει από κοινού. Δεν είμαι ικανοποιημένη με ένα σημείο. Το κείμενο αυτό αρχικά έφερε τον τίτλο Package Retail Information και κάποια protection scheme, αν δεν κάνω λάθος, και βλέπουμε τελικά ότι είναι απλώς ένα kid. Δηλαδή ανάμεσα στον τίτλο τον οποίο φέρει και το περιεχόμενο το οποίο πραγματικά έχει, υπάρχει μια κάποια διαφορά. Ουσιαστικά βγαίνουμε χαμένοι. Θέλω λοιπόν, ελπίζω ότι με τη δική μας την κοινωνιστική εργασία θα καταφέρουμε να εμπλουτίσουμε εκ νέου το κείμενο αυτό. Και συγκεκριμένα θα πρέπει να καταφέρνουμε να ενημερώνουμε για κάποια προϊόντα και να τα πιστοποιούμε προτού αυτά βγούνε στην αγορά και να δούμε πώς θα καταφέρουμε να διευθυντήσουμε και το ζήτημα του επόπτη, το οποίο μας απασχολεί πολύ συχνά. Ξέρω ότι τα ζητήματα αυτά απασχολούν πολλές φορές α, πολλές χώρες. Πρέπει λοιπόν να τα διευθετήσουμε από κοινού. Όσον αφορά το, τη γεφύρωση αυτή που θα πρέπει να γίνει με το ΟΣΕΚΑ, το ζήτημα αυτό το έχω αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν. Υπάρχουν στοιχεία στα πλαίσια του ΟΣΕΚΑ, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρουμε και στο κείμενο αυτό, όσον αφορά το ζήτημα της ευθύνης, για παράδειγμα. Νομίζω ότι ε, υπάρχουν κάποιες εξωτερικές ομάδες οι οποίες ασκούν πίεση θα πρέπει να δούμε πραγματικά, θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση όσον αφορά τα κριτήρια κινδύνου. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα αναφέρατε οι περισσότεροι. Ξέρω ότι δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο τι έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά να δούμε και τι μας περιμένει στο μέλλον. Θα πρέπει να γνωρίζουμε επίσης και ποιος είναι ο, ρίσκος, ε, συγγνώμη, ο κίνδυνος ρευστότητας. Θα πρέπει και αυτό να αναφέρεται στο νομοθετικό αυτό πακέτο. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα των συντάξεων, και εγώ ασχολήθηκα με το ζήτημα αυτό. Στα πλαίσια του ΠΡΥΠΣ υπάρχουν κάποια σταξιδωτικά προϊόντα τα οποία καλύπτονται. Τα ιδιωτικά σταξιδωτικά όμως μία δεν καλύπτονται. Δίστασα λοιπόν στην αρχή για το τι θα έπρεπε να κάνουμε και η άποψή μου είναι ότι δεν θα πρέπει να κινηθούμε στην κατεύθυνση αυτή για πολλούς λόγους. Καταρχάς, γιατί θα πρέπει να επιτευχθεί μια ισορροπία στο κείμενο και δεν θα πετύχουμε την ισορροπία αυτή αν εντάξουμε στο κείμενο τα pension funds, τα ιδιωτικά συνταξιδοτικά ταμεία. Καταλαβαίνετε ότι το κείμενο θα είναι ιδιαίτερα ανισόρροπο. Ενδεχομένως το κείμενο να αρχίσει να ασχολείται μόνο με τα ιδιωτικά στα ταμεία, όλες οι διατάξεις να επικεντρώνται στα προϊόντα αυτά και να μην καταφέρουμε να καλύψουμε ισότιμα τα υπόλοιπα επενδυτικά προϊόντα. Ελπίζω ότι ε, η αναθεώρηση του ΠΡΙΠΣ θα μας επιτρέψει να καλύψουμε και τα προϊόντα αυτά, δηλαδή τα ιδιωτικά συντοξιστικά ταμεία. Χαίρομαι που υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της φορολογίας και του φορολογικού καθεστώτος των επενδυτικών προϊόντων. Θα είναι δύσκολο να το κάνουμε αυτό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να επιμείνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος παράγει το προϊόν, ποιος μου διαθέτει το προϊόν και επομένως πρέπει να έχω τις απαραίτητες πληροφορίες για το προϊόν αυτό. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες ε, των ε, αρχών επιτήρησης, το ζήτημα αυτό το κάλυψα ποιες συνθήκες θα πρέπει να υπάρχουν όσον αφορά την απόσυρση συγκεκριμένων προϊόντων, ποιες πληροφορίες θα πρέπει να υπάρχουν προτού τα προϊόντα διατεθούν στην αγορά. Όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα, το κρατικό χρέος. Ναι, αναφέρθηκα στο κρατικό χρέος, αλλά αναφέρομαι κυρίως σε ομόλογα αν το ελληνικό χρέος μπορούσε να προταθεί στο ευρύτερο κοινό, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, αν υπήρχαν επιδυτικά προϊόντα τα οποία θα σχετίζονταν με το ελληνικό χρέος, τότε προφανώς θα πρέπει να συνοδεύονται τα προϊόντα αυτά με τις απαραίτητες πληροφορίες. Θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζει ο επενδυτής, ο μικροεπενδυτής, που επενδύει, ακόμα και συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Νομίζω πάντως ότι το δημόσιο χρέος δεν αγοράζεται πλέον τόσο πολύ από μικροεπενδυτές, εκτός και αν έχουμε τίποτα τελευταίες εξελίξεις, τις οποίες δεν γνωρίζω. Πάντως νομίζω ότι δεν ήθιστε πλέον η επιλογή αυτού του προϊόντος από τους μικροεπενδυτές. Όσον αφορά την πλήρη διαφάνεια για τα τέλη και το κόστος, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε εδώ πέρα την συζήτηση που είχαμε κάνει στα πλαίσια του MIFID. Τέλος, συμφωνώ και με τον Φίλιπ Λαμπέρ, ο οποίος είχε, μάλλον είναι στην αίθουσα, ναι, τον βλέπω. Όντως, θα πρέπει να προβλέπετε ότι ε, ο καταναλωτής, ο επενδυτής έχει διαβάσει τις πληροφορίες αυτές και μάλιστα να πιστοποιείται ότι όντως τις αποδέχεται. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα διαβάσει βέβαια όλα αυτά τα κείμενα, αλλά μη τι άλλο καλύπτουμε και την προϋπόθεση αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως έχουμε κάνει με άλλα προϊόντα. Δηλαδή να φαίνεται κάπου ότι ο επενδυτής πιστοποιείται ότι έχει ενημερωθεί για τα προϊόντα αυτά. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και την νομική υπηρεσία που με βοήθησαν. Ευχαριστούμε πολύ, λαμβάνοντα υπόψη και άλλες συζητήσεις που έχουμε κάνει για την επίλυση των κρίσεων. Ενδεχομένως και εδώ θα πρέπει να δούμε ποια κριτήρια ακριβώς μπορούμε να εντάξουμε στα προϊόντα αυτά. Κάνουμε λοιπόν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Στις 28 Νοεμβρίου θα έχουμε το σχέδιο έκθεσης. Στις 10 Νοεμβρίου θα είναι η προθεσμία καταβολής των τροπολογιών. Στις 21 Ιανουαρίου θα εξετάσουμε αυτές τις τροπολογίες. Στις 20 Μαρτίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και η έκθεση αυτή θα πάει στην Ολομέλεια του Απριλίου. Αυτό είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας προχωρήσουμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Θα δώσω την Προεδρία στον Αντιπρόεδρό μας. Σας ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης που είναι η οδηγία για την διαμεσολάβηση στα θέματα ασφαλιών, η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και όπως ξέρετε ο κύριος Λάγκεν είναι ο εισηγητής και στον οποίο θα δώσω αμέσως το λόγο. Βέρνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί με τη Γραμματεία έχουμε συντάξει ένα έγγραφο εργασίας στις 16 Οκτωβρίου σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν για τη διαμεσολάβηση στα ασφαλιστικά θέματα. Σε τέσσερις περίπου σελίδες έχουμε προσπαθήσει να καλύψουμε τα βασικότερα στοιχεία της πρότασης της Κομισιόν. Δεν είναι η οριστική μας αξιολόγηση βέβαια, είναι απλώς ε, ένας κατάλογος περισσότερο των εκκρεμών θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η διαδικασία αυτή θα κρατήσει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα οριστικό κείμενο και ευχαριστώ τη Γραμματεία για την υποστήριξή της. Το σχέδιο αυτό που έχετε ενώπιόν σας, το εγγραφό εργασία, είναι τμήμα της ε, γενικής διαδικασίας ρύθμισης που πρέπει να καλύψει και τα ασφαλιστικά προϊόντα και φυσικά στοχεύει στο να εξασφαλίσει και ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για τα προϊόντα της, ε, ασφαλιστικού χαρακτήρα και στη βελτίωση επίσης αποσκοπή της προστασίας των καταναλωτών και επομένως βρισκόμαστε σε συνεργασία με την Επιτροπή ΙΜΚΟ η οποία είναι και αυτή αρμόδια για τα θέματα αυτά εγώ πιστεύω όμως ότι η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να παραμείνει αρμόδια επί της ε, ουσίας, γιατί εμείς έχουμε την υποχρέωση να εκπονήσουμε ένα συνολικό πακέτο για τα θέματα αυτά. Είναι σαφές ότι η ΙΜΚΟ, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για το θέμα αυτό και ιδίως για το θέμα των προϊόντων που έχουν να κάνουν όμως με την ασφάλεια ζωής και τα προϊόντα μακροχρόνιου χαρακτήρα. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι στη δική μας αρμοδιότητα. Δεν χρειάζεται να εξάρω τη σημασία του ασφαλιστικού τομέα. Έχουμε περίπου ένα εκατομμύριο μεσίτες ασφαλιστικών ε, συμβολέων. Ένα μεγάλο μέρος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η διαμεσολάβηση είναι ένα σημαντικός επιχειρηματικός τομέας που παίζει μεγάλο ρόλο στον ε, τομέα ασφάλειας ε, πάνω από 90% σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ισπανία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο κτλ. Είναι λοιπόν ο τομέας αυτός πάρα πολύ σημαντικός, ο τομέας της διαμεσολάβησης. Μειώνει το κόστος αναζήτησης για τον ε, καταναλωτή, βοηθούν ιδιαίτερα στο να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες συμβάσεων για, την, ε, για τα ασφαλιστικά συμβόλαια, μειώνουν τον κίνδυνο <clears throat> για τους καταναλωτές και βοηθούν πάντα τους καταναλωτές να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν με τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες και την γραφειοκρατία που πρέπει να αντιμετωπίσουν για τη σύναψη ή την κατάργηση των συμβολέων αυτών. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τη βάση της ε, ήδη υπάρχουσας οδηγίας για τη διαμεσολάβηση η οποία είχε, από, είχε εγκριθεί στις 2 Νοεμβρίου 2002 έχει, είχε την πρόθεση να υπάρξει μια ε, επανεξέταση αυτής της οδηγίας επί και βάση της εμπειρίας και σε γενικές γραμμές. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια ε, ελάχιστη εναρμόνιση για τα θέματα αυτά, χωρίς φυσικά να μπορέσει να προκύψει μια πλήρης εναρμόνιση και να απαιτηθεί μια πλήρης εναρμόνιση για την αρκετά ετερόκλητη αγορά διαμεσολάβησης προϊόντων. Επίσης τα θέματα που αφορούν τα πρίψη αυτά τα ασφαλιστικά προϊόντα θα πρέπει να αποτελέσουν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο αυτή τη οδηγία. Το γεγονό λοιπόν ότι έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο διαμεσολαβητέ στον ασφαλιστικό τομέα θα πρέπει να μας ε, αποτρέψει από το να προχωρήσουμε σε υπερβολική ε, ρύθμιση η οποία δεν θα βοηθήσει ούτε τους καταναλωτές ούτε την αποτελεσματικότητα της αγοράς διαμεσολάβησης. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρξει υπερβολικό διοικητικό κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα πρέπει να περιορίσουμε και την ε, ρύθμιση για τα πολύπλοκα αυτά προϊόντα. Η Κομισιόν σε μεγάλο βαθμό έχει τηρήσει αυτό το κανόνα, σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια δεν το τηρεί απόλυτα. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το, καταρχήν το πεδίο εφαρμογής, όπου η Κομισιόν στο άρθρο 1 προτείνει να διευρυνθεί η σφαίρα εφαρμογής στους ασφαλιστές και επανασφαλιστές που δεν έχουν ε, συμμετοχή ενδιαμέσων και επίσης στους ε, εκτιμητές των ε, αξιώσεων κτλ. Είναι όλα αυτά στοιχεία για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε κατά πόσο η συμμετοχή των εκτιμητών ζημιών παραγωγή χάρη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτοί οι οποίοι παρέχουν τεχνικές εμπειρογνωμοσύνης κατά πόσο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής αυτής της ε, έκθεσης. Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή δεν συμβουλεύει να ληφθούν υπόψη και οι εκτιμητές αξιώσεων. Επίσης, υπάρχει το θέμα της συμπερίληψης ασφαλιών ταξιδίου, παραδείγματος χάρη που έχει μεγάλο όγκο με συνολικό, συνολική συμμετοχή στον ασφαλιστικό τομέα περιορισμένη μεν, αλλά κάθε χρόνο έχουμε 140 τέτοιες ασφαλίσεις ταξιδίων οι οποίες είναι παράπλευρα προϊόντα μιας αγοράς χάρη, ταξιδιωτικών πακέτων. Αυτά λοιπόν είναι περιορισμένα σε ύψος, πολλές φορές παίρνει κανείς ένα προϊόν το οποίο καλύπτει τα ταξίδια για ένα ολόκληρο χρόνο, είναι περιορισμένα τα, το συνολικό, συνολικός αυτών των προϊόντων. Μπορούν να παραμείνουν λοιπόν σε εξαίρεση όλα αυτά τα προϊόντα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τους καταναλωτές. Αλλά η συμπερίληψη σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πρόσθετη συμμετοχή διαμεσολαβητή για τα γραφεία ταξιδίων αν συμπεριληφθούν αυτά τα, αυτές οι μορφές ασφάλεια, ή μπορεί να απαιτηθεί από τους υπαλλήλους των γραφείων ταξιδίων να έχουν ιδιαίτερα προσόντα. Κάποιο ο οποίο κάνει ένα ταξίδι μπορεί να ασφαλιστεί για τον κίνδυνο να υπάρξει πρόβλημα για, την, για τον επαναπατρισμό του. Αυτό είναι συνήθω ένα μικρό ποσό και μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα όσα έχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν επίση τα θέματα του leasing αυτοκινήτων. Είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και <clears throat> υπάρχει πολλές φορές μια τεράστια διαφορά σε ρυθμίσεις. Κανείς δεν ξέρει όταν νοικιάζει ένα αυτοκίνητο τι ακριβώς περιλαμβάνεται σε αυτήν την πρόσθετη ασφάλιση. υπάρχουν και τα θέματα των πρόσθετων ασφαλιών που θα πρέπει να είναι διάφανα προς τον καταναλωτή πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό τονίζω ότι θα πρέπει οι συμφωνίες leasing όταν συνδέονται με πρόσθετες παροχές ασφάλειας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται χωριστά. Επανέρχομαι πάλι στο τομέα Αυτά για το τομέα εφαρμογής. Το άλλο είναι η διαδικασία εγγραφής, στα άρθρα 2, 3 και 4 και η απλοποιημένη διαδικασία δήλωσης. Εδώ το ερώτημα είναι ποιος θα πρέπει να καταγράφεται σε μητρό. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες στα κράτη-μέλη. Και το ερώτημα είναι αν με την διεύρυνση του τομέα εφαρμογής για άλλους φορείς διαμεσολάβησης θα πρέπει όλοι αυτοί να υπόκεινται σε υποχρέωση καταγραφής. Η Κομισιόν δεν το ζήτησε αυτό, αλλά ορισμένε ενώσει έχουν επιμείνει ότι πρέπει να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία. Εγώ πιστεύω όμως ότι δεν είναι απαραίτητη μια τέτοια νέα καταγραφή εάν έχουν ε, ήδη μια δραστηριότητα. Οι επαγγελματικοί η Κομισιόν θέλει να διευκολύνει και να απλοποιήσει τη διαδικασία για αυτούς οι οποίοι ε, ασχολούνται με ταξιδιωτικά πρακτορία και ενοικίαση αυτοκινήτων και εκεί δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω γραφειοκρατία. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μιας απλοποιημένης ε, διαδικασίας. Ένα τρίτο σημείο είναι η περαιτέρω κατάρτιση και η πρόσθετη κατάρτιση των διαμεσολαβητών στον ασφαλιστικό τομέα. Εδώ νομίζω ότι έχει νόημα να υπάρχει μια σειρά υποχρεώσεων 200 ώρες σε 5 χρόνια παραδείγματος χάρη σε σχέση με τα νέα προϊόντα, τις νέες νομικές διατάξεις κτλ. Μία εβδομάδα το μήνα κατά κάποιο τρόπο, ε, κατά μέσον όρο 40 ώρες την, ε, το χρόνο. Υπάρχουν προτάσεις από διάφορες ενώσεις, όλα αυτά είναι εφικτά. Το θέμα είναι πώς θα γίνεται και πού θα γίνεται αυτή η εκπαίδευση. Θα πρέπει να είναι κάποιος ιδιαίτερος φορέας κατάρτισης. Θα πρέπει οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες να αναλάβουν την πιστοποίηση τέτοιων φορέων κτλ. Νομίζω ότι για μένα είναι πολύ σημαντικό ο τομέα αυτό τη κατάρτιση, γιατί έρχονται τόσα πολλά καινούργια προϊόντα στην αγορά, ιδίω για μακροπρόθεσμα ασφαλιστικά συμβόλαια, που θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα για αυτό το θέμα. Περνάω στο τέταρτο σημείο, στο άρθρο 17, δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων και διαφάνεια. Και εδώ υπάρχει μια πλειάδα προτάσεων και υπάρχει και έντονη συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να συμπεριληφθούν διατάξεις αυτού του είδους, όπως έχουμε κάνει και στα πλαίσια της οδηγίας MIFID, πώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί λοιπόν η διαφάνεια και η έλλειψη συγκρούσεων Ε, προτείνεται να υπάρχουν και εδώ επεκτάσεις αυτών των προτάσεων ε, που ήδη ισχύουν. Εγώ θεωρώ ότι αυτό όμως θα οδηγήσει σε μια μορφή στρέβλωσης. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να προσπαθήσουμε να πετύχουμε την προστασία των καταναλωτών με μέτρα τα οποία θα είναι αδιαφανή αν έχουμε παραγωγή χάρη μια συμφωνία μέσω του ίντερνετ η οποία προτείνει ένα μακροχρόνιο προϊόν όπως μια ασφόλη, ασφάλεια ζωής όταν πρόκειται λοιπόν για καταναλωτές οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν τις απαραίτητες ε, συμβουλές και οι συμβουλές αυτές παρέχονται από τον ασφαλιστή αλλά σε κόστος, με κόστος του καταναλωτή, αυτή η διαδικασία δεν έχει καμία διαφάνεια και δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και το γεγονός ότι οι πολίτες δεν θέλουν να υπάρχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις θα πρέπει να μας οδηγήσει να αποφύγουμε μια τέτοια αντιμετώπιση. Ακόμα και οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών στην Ευρώπη ε, θα πρέπει να το αναγνωρίσουν αυτό. Μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη, αλλά εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει να ακούσουμε του εμπειρογνώμονες και όχι τις ενώσεις των καταναλωτών. Επίσης υπάρχει το θέμα της διαφάνειας της ε, αποκάλυψης, της πλήρους αποκάλυψης των προσθέτων τελών και του συνολικού κόστου αυτών των προϊόντων η δική μου εντύπωση δεν είναι ότι το βρετανικό σύστημα, το σύστημα on request, δηλαδή μόνο με την ε, αίτηση του καταναλωτή θα πρέπει να λειτουργεί. Αυτό δεν έχει <clears throat> αποδείξει την αξία του στο παρελθόν. Υπάρχουν ε, άλλες χώρες όπου η <clears throat> οι ασφαλιστές έχουν νομικές υποχρεώσεις για να δίνουν πληροφορίε. Η παρουσίαση λοιπόν όλων αυτών των στοιχείων που ενδιαφέρουν τον καταναλωτή μόνο με αίτηση του καταναλωτή ε, πολλές φορές δεν δίνει τα απαραίτητα αποτελέσματα. Υπάρχουν και τεχνικές ε, δυσκολίες πολλές φορές στην εκτίμηση των διαφορών στοιχείων. Η πρότασή μου είναι να αναφέρεται η φύση και το ύψος του πρόσθετου κόστους ώστε να υπάρχει αυτή η πληροφόρηση του καταναλωτή. Θα πρέπει όμως και αυτό να το συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορεί να τροποποιηθεί η πρόταση της Κομισιόν για τα θέματα αυτά και εγώ θα προτιμούσα να αφήσουμε την αυτορύθμιση στα κράτη-μέλη για όλα αυτά τα θέματα. Στη συνέχεια έχουμε τα λεγόμενα προϊόντα επενδύσεων σε επίπεδο ε, ασφαλιστικών προϊόντων που συνδέονται και με την οδηγία MIFID. Εδώ λοιπόν ε, αυτό που παίζει ρόλο είναι πώς θα αντιμετωπίζονται τα προϊόντα αυτά κατά πόσον δηλαδή θα πρέπει να συγκρίνονται με αμυγός επενδυτικά προϊόντα, άρα δηλαδή υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς ή μήπως θα πρέπει ως προϊόντα ασφαλιστικών επενδύσεων να αντιμετωπίζονται διαφορετικά, δηλαδή να είναι αντικείμενο συναλλαγών ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εδώ υπάρχουν διάφορες δυνατότητες, μπορεί να υπάρξει και κάποια λύση, δηλαδή προϊόντα τα οποία ε, δεσμεύονται με ταμεία, υπάγονται στην MIFID μόνο εφόσον δεν υπάρχει το κατώτατο χρονικό διάστημα και υπάγονται όλα τα άλλα που είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας. Τα ε, επενδυτικά προϊόντα μεγάλης διάρκειας, ακόμα και αν δεσμεύονται με ταμεία, αυτά υπάγονται ε, στην οδηγία περί ασφαλιών και όλα τα άλλα στη MIFID. Πρέπει βέβαια να το συζητήσουμε και αυτό. Και υπάρχουν παραδείγματα τα οποία ε, από άλλες χώρες και από τη Φινλανδία που δείχνουν ότι αν είναι κανείς ε, άκαμπτος στο θέμα αυτό, ας πούμε και στο σύστημα των ε, αμοιβών, δηλαδή ότι μπορεί η υπαρχή συμβουλών να γίνεται μόνο επαμοιβή, αυτομάτως θα προκύψει, υπάρχει φόβος ότι θα προκύψει κακή ενημέρωση των πολιτών. Στη Φιλανδία που υπήρξε αυτό, τελικά μειώθηκαν τα ασφαλιστικά συμβόλαια αντί να αυξηθούν. Γιατί πριν πάει κανείς να πληρώσει για να συμβουλευτεί, να πάρει συμβουλές, το βήμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και έτσι κι αλλιώς και τα προϊόντα είναι ε, δύσκολα συγκρίσιμα. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλύτερο να υπάρχει απόλυτη ε, διαφάνεια των λογαριασμών των ασφαλιστικών εταιριών έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να ξέρουν τι παρακρατούν οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες για παροχή συμβουλών. Πάμε τώρα στις ε, κατεξουσιδότηση πράξης. Εδώ παίζει ρόλο η εναρμόνιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εδώ και πάλι προτείνει μια σειρά κατεξουσιοδότηση πράξεων, να οριστούν ε, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Όλα αυτά που αναφέρει λοιπόν η Κομισιόν στο αίτημά της για κατεξουσιοδότηση πράξης. Όλα αυτά επιθυμεί να τα ρυθμίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς κοινοβουλευτική συμμετοχή. Έχοντας λοιπόν κατά νου ε, τη ρύθμιση περί αποζημίωσης ε, ζημιών, θέλει τώρα εδώ η Κομισιόν από το παρατηράκι να εισάγει την ίδια ρύθμιση. Αν όμως το δεχτεί κανείς αυτό απλά, όπως το προτείνει η Κομισιόν, τελικά αυτό ε, θα οδηγήσει σε μία μέγιστη και όχι ελάσσονα εναρμόνιση και με αυτήν συνδέονται μία σειρά γραφειοκρατικών ρυθμίσεων ακόμα και αν το προϊόν αυτό πράγματι ε, συνδέεται με κάποιον προστατευτισμό. Εγώ όμως λέω να μην υπάρξει εδώ ελάχιστη de minimis ρύθμιση και να, δώσουμε την, ε, να, να τις υπόλοιπε αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Γίνεται, υπάρχουν πολλές έρευνες σχετικά με αυτή την οδηγία, ασφαλιστική οδηγία. Εμείς όμως εδώ στο Κοινοβούλιο εξαιρουμένων των θεμάτων που παίζουν ρόλο με τα μακροχρόνια επενδυτικά προϊόντα. Νομίζω ότι μπορούμε γρήγορα, σύντομα μάλλον, να βρούμε μια λύση και το χρονικό διάστημα σημαίνει ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου πρέπει να έχει κατατεθεί και σχέδιο έκθεσης, θα το καταθέσω εγώ ε, και η γραμματεία μου, 17 και 18 Δεκεμβρίου θα έχουμε τη μετάφραση. Πριν από τα Χριστούγεννα θα μπορούμε μπορούμε να κάνουμε μία πρώτη συζήτηση και η προθεσμία ε, τροπολογιών θα είναι αμέσω μετά τον Ιανουάριο. Θα ε, ψηφίσουμε από αυτού στις 26 Ιανουαρίου εδώ στην Επιτροπή μας. Και πριν μπούμε στον Τρίλογο, ε, θα έλεγα η ψήφιση στην Ολομέλεια να γίνει τον Απρίλιο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λάγκεν. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την διευκρίνηση του ποιο θα έχει την αρμοδιότητα επί τη ύλη μεταξύ τη δική μα Επιτροπή και τη Επιτροπή ΙΜΚΟ. Δεν έχει ληφθεί ακόμα η απόφαση αυτή. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάντσε Περσέδο για τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάγκεν για το έγγραφο εργασία του. Νομίζω ότι είναι ένα έγγραφο το οποίο έχει αντικειμενικό χαρακτήρα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, μας αναφέρει τα βασικά προβλήματα και τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να διαλευκανθούν σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Έχει παρουσιάσει λοιπόν και με την παρέμβασή του όλα αυτά τα στοιχεία. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω τα οριστικά συμπεράσματα για όλα αυτά τα ζητήματα, απλώς θέλω να κάνω μερικά περιορισμένα σχόλια. Πιστεύω ότι η πρόταση αυτή της Κομισιόν είναι απαραίτητη εδώ και 10 χρόνια. Είχε διαρκέσει η λειτουργία της προηγούμενης οδηγίας για τα ασφαλιστικά προϊόντα. Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια είναι σαφές ότι έχουν γίνει πολλά γεγονότα και ούτως ή άλλως η τρέχουσα οδηγία προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2015. Γι' αυτό είναι πολύ σωστή η πρωτοβουλία αυτή της Κομισιόν. Και ουσιαστικά με την οδηγία αυτή υλοποιούμε δεσμεύσει που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των G20 και είναι πολύ απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ισότητα ανταγωνισμού για τα ασφαλιστικά θέματα. Τα θέματα του ανταγωνισμού φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικά όπως θα τονίσει και η Επιτροπή ΙΜΚΟ για όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαμεσολάβηση είναι απαραίτητο να υπάρχουν κανόνε που θα εξασφαλίσουν τον θεμητό ανταγωνισμό στον τομέα αυτό. Είναι επίση όμω απαραίτητο να βελτιώσουμε και την προστασία των καταναλωτών και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την Εκτελεστική Επιτροπή. Είναι και ένα στοιχείο τη πολιτική ανταγωνισμού. Και επίση είναι απαραίτητο να προωθήσουμε την μεγαλύτερη ολοκλήρωση τη αγορά ασφαλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο θα οδηγήσει και σε οικονομικό όφελος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για μια ρύθμιση η οποία θα οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα <clears throat> και αξιοπιστία της αγοράς. Υπάρχουν φυσικά μια, υπάρχει μια πλειάδα σημαντικών και ευαίσθητων θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια, την ανταγωνιστικότητα, την πληροφόρηση, τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι οικουμενική αυτή η ρύθμιση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει η σωστή αντιμετώπιση των θέματων ανταγωνισμού, που δεν θα είναι γεγονός αν παραμείνουν εκτός του, της σφαίρας εφαρμογής τομή. τομής. Η οικουμενικότητα όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένα στοιχεία, όπως είναι η πολυπλοκότητα του τομέα των ασφαλιών. Υπάρχουν ε, τα ασφαλιστικά συμβόλαια του κλάδου ζωής, του, των υπολείπων κλάδων, πρέπει σε κάθε περίπτωση να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών, της ιδιαιτερότητες αυτών των προϊόντων και πολλές φορές συνδέονται τα με, με τα δε. Και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τελείως αυτόνομα όλες αυτές τις μορφές ασφαλιών. Πολλές φορές ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα ε, συν, συνάπτονται σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες ή άλλες αγορές. Παραδείγματος χάρη το συμβόλαιο για την ε, ασφάλεια ενός υπολογιστή όταν αγοράζει κανείς ένα προσωπικό υπολογιστή. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αποφύγουμε ότι στην προσπάθεια να ρυθμίσουμε τα πάντα θα καταλήξουμε σε αρνητικά αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να φρενάρουμε την υπερβολική ε, φιλοδοξία της νομοθεσίας για την καταγραφή των ε, διαμεσολαβητών, πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή εγγραφής αυτών και κάποια δήλωση από τη δική τους πλευρά για όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα αυτό. Είναι απαραίτητο επίσης να εξασφαλίσουμε τον επαγγελματικό χαρακτήρα των διαμεσολαβητών αυτών που θα πρέπει να το προωθήσουμε και επομένως όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις γνώσεις και την κατάρτισή τους θα πρέπει να τα εξάρουμε ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο και επίσης να λαβω υπόψη και την επαγγελματική τους διοντολογία. Και εδώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων με τις κατάλληλες λύσεις. Αυτά ήθελα λοιπόν να πω για τις επιμέρους ε, πτυχές. Έχουμε και άλλα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, παραδείγματος χάρη το θέμα των ε, ενυπόθηκων δανείων στεγαστικών δανείων κτλ. Όπου πολλές φορές υπάρχουν προϊόντα πακέτο τα οποία απολούνται τα συνδεόμενα προϊόντα λοιπόν αυτά τα οποία μπορεί κανείς να αγοράσει είτε από κοινού είτε χωριστά. Είναι κάτι σαν να πηγαίνει κανείς σε ένα εστιατόριο παραγωγικά και υπάρχει το μενού της ημέρας αλλά δεν μπορεί κανείς να ε, φάει κάτι αλακάτ. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να πάρει μόνο ένα συγκεκριμένο προϊόν, ότι πέραν του μενού της ημέρας μπορεί να φάει και κάτι διαφορετικό και να γίνεται μια αντίστοιχη αντιμετώπιση στον τομέα των ασφαλιών. Επίσης η διαμεσολάβηση πολλές φορές έχει και ιδιαίτερες πτυχές, όπως είναι η εκτίμηση και η παροχή συμβολών συμβουλών. Θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση μεταξύ της παροχής συμβουλών στα ασφαλιστικά προϊόντα και της προώθησης του μάρκετινγκ. Πρέπει να κρατήσουμε χωριστές αυτές τις ε, διαδικασίες, γιατί η παροχή συμβουλών δεν θα πρέπει να έχει σαν στόχο την βελτίωση της κερδοφορίας μιας επιχείρησης, αλλά να εξασφαλίσει τα συμφέροντα των καταναλωτών και εκεί επομένως θα πρέπει να υπάρχει μια πιο προσεκτική και αυστηρή ρύθμιση. Σημερίζουμε επίσης και αυτά τα οποία έχουν ελεχθεί ότι για τα επενδυτικά προϊόντα να εφαρμοστούν οι λύσεις που έχουμε εγκρίνει και σε άλλους τομείς για να μην υπάρχουν αντιφάσεις και διαφορετικές ρυθμίσεις, αλλά παράλληλα ο στόχος μας είναι εναρμόνιση θα πρέπει να είναι μια λογική εναρμόνιση. Δεν μπορούμε να εναρμονίσουμε τα πάντα. Το θέμα ε, προς τα ελάχιστα ή προς τα μέγιστα της εναρμόνισης δεν είναι το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό είναι να είναι συνεκτική αυτή η εναρμόνιση και να μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ κύριε Σάτσερ Πεσέδο. Από τους φιλελεύθερους ο κύριος Σμιτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστήσω και τον κύριο Λάγκεν για την εργασία που έχει κάνει. Συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία υπόθηκαν και στο κείμενο λέτε ότι χρειαζόμαστε μια πιο αυστηρή προστασία των επενδυτών. Και συμφωνούμε. Συμφωνούμε όλοι. Λέτε όμως και κάτι ακόμα. Ότι θα πρέπει να έχουμε καλά λειτουργούσες αγορές. Πολλές φορές η υπερβολική ρύθμιση δεν είναι επιθυμητή. Αυτό λέτε επίσης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε ακριβώς ποια είναι η αναλογικότητα των πράξεών μας. Κάνουμε όντως πράγματα τα οποία βοηθούν ή μπορεί να ταχθούν και κατά των ίδιων των καταναλωτών. Χαίρομαι πάρα πολύ που θίγεται πάντως το ζήτημα της αναλογικότητας της παρεμβολής μας. Στα πλαίσια του MIFID 2 ενό πολύπλοκου νομοθετήματο ασχοληθήκαμε με το ζήτημα αυτό και λέτε και εσεί πολύ σωστά ότι η εν λόγω νομοθετική πράξη θα πρέπει να συνάδει, να ευθυγραμμιστεί με το MIFID 2, αποφεύγοντα επικαλύψει. Αναφέρεστε επίση το ζήτημα τη ε, πλήρου ε, εναρμόνιση. Ζήτημα το οποίο μα απασχόλησε και στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ο καλύτερο τρόπο τελικά για να προχωρήσουμε. Συμφωνώ ότι υφίστανται προβλήματα στη λύση αυτή και αν τελικά ορισμένες χώρες θέλουν τουλάχιστον σε μια μεταβατική περίοδο να εφαρμόσουν πιο αυστηρούς κανόνες όπως έχουμε προβλέψει και στα πλαίσια του MIFID, τότε δεν μπορούμε να στερήσουμε από τις χώρες αυτές αυτή τη δυνατότητα. Όσον αφορά τώρα το πεδίο εφαρμογής, στα πλαίσια του MIFID προσπαθήσαμε να καλύψουμε κάποια από τα κενά τα οποία υπήρχαν, το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε και εδώ και να δούμε τελικά τι είναι συγκρίσιμο ανάμεσα στην πρόταση αυτή και το MIFID. Και εσύ είμαστε και προσεκτικοί, ας μην δημιουργήσουμε επικαλύψεις. Και υπάρχουν ε, πολλές διαφορετικές ε, ασφάλειες, πολλά διαφορετικά είδη ασφάλειας και ασφαλιστικών προϊόντων τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε. Να λάβουμε δηλαδή υπόψη και τις ιδιαιτερότητές τους. Αναφερθήκαμε επίσης και στο PRIPS, συνάδουν τα όσα είπαμε για το PRIPS με τα όσα λέμε εδώ πέρα. Όσον αφορά τα προϊόντα εγγύησης των καταθέσεων, και αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο ορισμό για τις συμβουλές, για την παροχή των συμβουλών. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και μας απασχόλησε και στα πλαίσια του MIFID. Και υπάρχει και το γενικό ζήτημα που έχει να κάνει με την διαφάνεια. Στα πλαίσια του μύθιτ είχαμε δει ότι υπήρχαν ορισμένες χώρες οι οποίες ε, μπορούσαν να απαγορεύσουν κάποια προϊόντα. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το να επιτρέψουμε να δημιουργηθεί ένα μη ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού. Δηλαδή να υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές, τόσο μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχει μία κάποια παραπλανητική πώληση των προϊόντων αυτών. Πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες και όταν λέω να τους προστατεύσουμε ενώ να τους δώσουμε τη σωστή ενημέρωση ως φιλελεύθερος καταλαβαίνετε ότι θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι ιδεοντολογικοί κανόνες, οι κανόνες συμπεριφοράς που κατά καιρού εγκρίνουμε, θεωρώ ότι δεν αρκούν πολλές φορές. και ενδεχομένω να πρέπει κατά καιρού να χρησιμοποιούμε και πιο αυστηρούς κανονισμούς ή ακόμα και απαγορεύσεις. Πάντως, τα όσα προβλέπονται στο MIFID θα μπορούσαν να εφαρμόζονται και συγκεκριμένη περίπτωση, Ενδεχομένω να τα αναφέρουμε στα εκτιμώντα τη έκθεση. Όσον αφορά τώρα την κατάρτιση, νομίζω ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό, το βλέπετε και στο έγγραφό σας. Η κατάρτιση και γενικότερη εκπαίδευση είναι δύο πολύ σημαντικά ζητήματα και εγώ είμαι σαφώ υπέρ τους. Πολλές φορές μας λένε ότι τα προβλεπόμενα προγράμματα δεν αρκούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να λέμε ότι η σωστή κατάρτιση και εκπαίδευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η σωστή κατάρτιση όσων πουλάνε τα προϊόντα αυτά, είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για να καταλήξουμε τελικά σε μια αγορά η οποία θα λειτουργεί σωστά. Νομίζω ότι στα σημεία αυτά θα καταφέρουμε να καταλήξουμε πραγματικά σε μια σημαντική συνένεση. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει κάποιο ε, τον λόγο για του πράσινους, ο κύριος Φιλίπ Λαμπέγα. Βλέπω ότι μου δίνετε πάρα πολλέ φορέ το λόγο σήμερα. Θα ήθελα να αντιδράσω σε αυτά που είπε όλε. Νομίζω ότι η προσέγγισή σου είναι πολύ λογική. Θέλουμε ο επενδυτής αλλά και ο να προστατευτούν. Θέλουμε μια αγορά που να λειτουργεί σωστά, θέλουμε να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, αλλά δεν θέλουμε, τουλάχιστον εγώ έτσι το καταλαβαίνω, να τον απαλλάξουμε εντελώ από τις ευθύνες του. Θα πρέπει δηλαδή ο καταναλωτής να λειτουργεί υπεύθυνα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν τόσα πολλά Τόσε πολλέ προστατευτικέ δικλείδε, ώστε τελικά ο καταναλωτή να αποποιείται των υποχρεώσεών του και τη ευθύνη του. Συμφωνώ λοιπόν με αυτή την ισοσκελισμένη, την ισορροπημένη προσέγγιση την οποία πρότεινε. Και εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος με, τα με τις απαγορεύσεις οι οποίες προβλέπονται στα πλαίσια του MIFID. Συμφωνώ με την ευελιξία την οποία θέλεις να προσδώσεις στο συγκεκριμένο νομοθέτημα. Είναι πάντως δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην ευθύνη και την προστασία. Κάποιες ε, προτάσεις να κάνω κι εγώ, με τι συμφωνούμε, τι θέλουμε να δυναμώσουμε, τι απουσιάζει από το κείμενο και πρέπει να προστεθεί. Συμφωνούμε με το πεδίο εφαρμογή τη ε, πρόταση. Όλες οι διατάξεις που έχουν να κάνουν με τις απαραίτητες γνώσεις για το διαμεσολαβητή είναι πολύ σωστές. Συμφωνούμε επίσης ότι αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι κανόνες ή αν δεν τηρούν οι απαραίτητοι κανόνες πρέπει να προβλέπονται κυρώσεις. Κανόνες χωρίς κυρώσεις ουσιαστικά δεν λειτουργούν στην πράξη, είναι μόνο θεωρητικοί. Συμφωνούμε επίση ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ποιότητα τη παρεχόμενη συμβουλή. Αυτά είναι τα σημεία από των οποία συμφωνούμε. Ζητήματα τα οποία πρέπει να δυναμώσουμε τώρα. Όπως και σε προηγούμενες συζητήσεις για το PRIPS, έτσι και εδώ, για ποιο λόγο στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι εξοδικαστικές διευθετήσεις δεν είναι δεσμευτικές. Για ποιο λόγο προβλέπετε κάτι τέτοιο, θέλουμε να το καταλάβουμε αυτό και θέλουμε ουσιαστικά να αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα αυτές οι διευθετήσεις. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της διαφάνειας, χρειαζόμαστε και εδώ πέρα ένα KID τελικά, δηλαδή κάποια βασικά έγγραφα ενημέρωση που θα δίνουν βασικές πληροφορίες του καταναλωτή και θα πρέπει βέβαια να υπάρχει μία απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά τις πληροφορίες αυτές και θα πρέπει επίσης να εμπεριέχονται και κάποια άλλα στοιχεία στην πρόταση αυτή τα οποία δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Θέλουμε να γνωρίζουμε ποια είναι η συνολική απόδοση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, αν πρόκειται για παράδειγμα για μια ασφάλεια ζωής και θα θέλουμε τελικά να γνωρίζουμε ποιο είναι το πραγματικό όφελος για το καταναλωτή αφού αφαιρεθούν όλα τα τέλη και όλα τα κόστη. Άλλες πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν είναι κάποιοι βασικοί δείκτες όσον αφορά τις πληρωμές για αποζημιώσεις ή για καθυστερούμενες αποζημιώσεις. Ξέρετε ότι πολλές φορές οι καταναλωτές είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι όταν βλέπουν ότι τελικά υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάνουν ένα αίτημα αποζημίωση μόνο και μόνο για να καλύψουν ότι τελικά δεν καλύπτονται για το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα ή ότι πολλές φορές καταφέρνουν να αποκομίσουν μια αποζημίωση αλλά μετά από πολλά χρόνια θα ήταν πολύ θετικό να έχουμε κάποια στατιστικά δεδομένα τα οποία να μας καταδεικνύουν τελικά πόσος χρόνος απαιτείται προκειμένου να αποπληρωθεί, να χορηγηθεί μια αποζημίωση στον καταναλωτή. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε επίση και ποιε είναι οι δικαστικέ προσφυγές που έχουν γίνει από καταναλωτές προ ασφαλιστικέ εταιρείε. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα. Όσον αφορά τώρα κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει κάπως να προσαρμοστούν, υπάρχει ένας ορισμός που αναφέρεται στον επαγγελματία καταναλωτή. Είναι σημαντικός ο ορισμός αυτός, γιατί ο καταναλωτής αυτός δεν χρειάζεται την ενημέρωση, της πληροφορίες που προβλέπονται στο κείμενο όσα λέγονται εδώ πέρα στο κείμενο αναφέρονται σε εταιρεία με ισολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ και δίνει επίσης και κάποια άλλα αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να καθοριστεί ο επαγγελματικός καταναλωτής. Αν συγκρίνουμε τον ορισμό αυτό με τον ορισμό που χρησιμοποιείται στη MIFID βλέπουμε ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να, θεωρεί, να θεωρεί ότι κάποιες επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν δικαιούνται να έχουν όλη αυτή την πλήρη ενημέρωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ορισμούς οι οποίοι να συνάδουν. Να έχουμε τον ορισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο κείμενο αυτό και ουσιαστικά αυτός ο ορισμός να αντιστοιχεί στο λεγόμενο επαγγελματικό επαγγελματία καταναλωτή. Και για λόγους συγκρισιμότητας σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει να έχουμε κοινού κανόνες, επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε και κοινού ορισμούς. Αν τώρα υπάρχουν κέρυοι λόγοι του τους οποίους εδώ πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας διαφορετικός ορισμός, τότε θα ήθελα να γνωρίζω ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό που έχουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο νομοθέτημα αυτό. Άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να δυναμωθούν στο κείμενο περισσότεροι κανόνες όσον αφορά τους διαμεσολαβητές οι οποίοι μεσολαβούν ανάμεσα στην ασφαλιστική εταιρεία και τον τελικό καταναλωτή. Μεγαλύτερη σαφήνεια για τον ρόλο των διαμεσολαβητών αυτών και κάποια ελάχιστα πρότυπα για τη δραστηριότητά τους. Ενδεχομένως η ΑΙΟΠΑ θα μπορούσε να επιληφθεί των λεπτομεριών αυτών. Αυτά τα σχόλια είχα να κάνω εξ του Σβέν και προφανώς θα συνεργαστούμε επικοδομητικά μαζί σας για, το, για την πρόταση αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Λάμπερτ. Έχουμε μόνο έξι λεπτά και έχουμε τρεις ομιλητές. Σας παρακαλώ να παραμείνετε λοιπόν ο καθένας στα δύο λεπτά. Η Κέι. Και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Και εγώ μιλώ εξ ονόματος της κυρίας Φόξ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λάγκεν για το έργο του, για το έγγραφο μέχρι στιγμής. Και να υπογραμμίσω όλα αυτά τα σημεία τα οποία επεσήμανε ήδη. είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση όπως και στην οδηγία μυφή. Θέλουμε όλοι να καταλήξουμε σε κοινή προσέγγιση και σε κοινού ορισμούς που θα οδηγήσουν σε ένα ισόπεδο γήπεδο το οποίο δεν θα γέρνει προς μια και θα δίνει ισότιμη προστασία σε όλους τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στο βαθμό του δυνατό ότι υπάρχει συγκρισιμότητα όλων αυτών των προϊόντων και ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά. Αλλά μετά τις συζητήσεις που έχουμε δει στην MIFID, υπάρχει και η συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις σε διαφορετικές αγορές και σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Μπορεί να μην υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση η οποία θα γίνει δεκτή από όλους. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν και κάποιο περιθώριο για τις εθνικές ιδιαιτερότητες και όπως και στην περίπτωση της ΜΥΦΙΤ είναι σημαντικό να μπορούν τα κράτη-μέλη να παροτηρηθούν να λειτουργούν μέσα σε μια κοινή αγορά, αλλά να μην τους αποτρέπουν να έχουν ένα πιο στεναρό καθεστώς προστασία των καταναλωτών εάν το επιθυμούν ο εισηγητής τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει και μία διαφοροποίηση μεταξύ των ε, αιτήσεων ε, για σύντομες ε, για τις, για τις σύντομες ε, ε, ασφάλειες ίσως είναι λιγότερο σημαντικό να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα πληροφοριακά σε σχέση με το συνολικό κόστος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να έχουμε μια συγκροτησμότητα και να επιστούμε περισσότερη την προσοχή των ε, καταναλωτών στα συγκριτικά στοιχεία. Ελπίζουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη διαφάνεια η οποία θα είναι αναλογική στα χρήματα τα οποία εμπλέκονται και πιστεύω ότι θα θέλαμε να τονίσουμε ιδιαίτερα τη σημασία του άρθρου 13 σε σχέση με την ύπαρξη θεραπείας, και αποκατάσταση και να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι συμβατό με την οδηγία περί εναλλακτικών συστημάτων <clears throat> επίλυσης διαφορών. Η κυρία Στάιλερ που είναι η συγγήτρια της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ και εγώ είμαι η στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Χαιρετίζω ιδιαίτερα αυτή την έκθεση. Θα έχουμε μία ακρόαση στην Επιτροπή μας στις 26 Νοεμβρίου θα σας πληροφορήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχετε υπόψη ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από κοινού το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Εν κατακλείδη ξαναδίνουμε το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Λάγκεν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για όλα αυτά που μας είπατε και όλα αυτά τα σημείωσα, τα κατέγραψα και αν κάποιος ε, έχει κάποιες άλλες παρατηρήσεις παρακαλώ να μου τις ε, στείλει τις επόμενες ε, δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση μέχρι τώρα και θεωρώ ότι η ΙΜΚΟ με την ακρόασή τη θα συνεχίσει το έργο. Ευχαριστούμε. Όπως είπε ο κύριος η έκθεση θα εξεταστεί στις 17-18 ε, Δεκεμβρίου του έτους. Η προθεσμία είναι 24 Ιανουαρίου και η εξέταση των τροπολογιών θα λάβει χώρα στις 18 και 19 Φεβρουαρίου. Και η ψηφοφορία θα ψηφίσει η Επιτροπή στις 26 Μαρτίου του επόμενου έτους. Η ψηφοφορία ε, θα γίνει στην Ολομέλεια του Απριλίου του επόμενου έτους. Και τέλος, η Γραμματεία θέλει να ενημερώσει τα μέλη ότι η έκθεση του κ. Στολόγιαν ε, θα εξεταστεί σήμερα το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν, μετά τις, ε, τις, τις, τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Ευχαριστώ πολύ.